So, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχει περάσει η ώρα μα Αλλά ήμασταν και λίγοι εδώ, ήμασταν μόνοι μα σχεδόν. Τώρα ήρθαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Ροτ Μπέραντ και ο κύριο Σλούτερ από ό,τι βλέπω δεν έχουν ε, καμία διάθεση για τροποποίηση σημερινή σα διάταξη. Την εγκρίνουμε λοιπόν και προχωρούμε στις Ανακοινώσει. Στη διάθεσή σας είναι όλες οι γλώσσες με διερμηνία και τα κροατικά, πλην τη εστονική και τη μαλτεζική γλώσσα. Όλες οι άλλες mm. Δεν έχετε διερμηνία. Αγγλικά δεν ακούγονται. Mm. Τώρα εντάξει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή σας με τα κροατικά μαζί, εκτός από τα εστονικά και τα μαλτεζικά. για την έκθεση Γκλής. Θα γίνει μια ε, σύντομη δεύτερη ανάγνωση. προκειμένου να προλάβουμε την 1η Ιουλίου για να γίνει η, ενσωμάτωσή της στην ε, νομοθεσία και να προλάβουμε να έχουμε και την μετάφραση εγκαίρως για τους Κροάτες. Επίσης, 24 Απριλίου, δηλαδή σήμερα, έχουμε ένα workshop για τα νεογνά στο ASP 5G2 Βίλμοτ, βιλμοντ αλλες Πίτσερλε θα είναι οι συνάδελφοι που θα, λάβουν, που θα παρουσιάσουν ε, το workshop αυτό σήμερα όπως είπαμε από τη μία μέχρι τις 3 παρατέταρτο και μετά έχουμε και ε, φοιτητές εδώ από το Μαριάψ, Ινστιτούτο του Βρυξελών. Από τις 3 μέχρι τις 3.30 θα είναι μαζί μας. Έχουμε και 20 μέλη του προσωπικού που ήρθαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πέμπτη ανακοίνωση έχουμε ένα νέο συνάδελφο, τον κύριο Φράνκο Ουνάνη, στην Επιτροπή μας από τους μη εγγεγραμμένους. Τακτικό μέλος. Αυτά προς το παρόν για τις ανακοινώσεις μας. Και έτσι περνάω στα πρακτικά της 17ης-18ης η δεκεμβριου αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα εγκρίνουμε και προχωρούμε στην έκθεση της κυρίας Dagmar Rock ιατρικός εξοπλισμός, ιατροτεχνολογικά προϊόντα καλύτερα. Μια έκθεση που θα συζητήσουμε μαζί με την έκθεση του κυρίου Πέτερ Λίζε για την ε, in vitro, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά ε, προϊόντα. Ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Ροτβέραντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέψετε θα μιλήσω στα αγγλικά. Με τη συμπάθεια των διερμηνέων ελπίζω. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε μια συνάντηση με τους σκιώδες και θέλω να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής διότι είναι ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί, καθώ υπάρχει ένα πλαίσιο ήδη τα τελευταία 20 χρόνια και θεωρώ ότι θέλω να πω ότι το καλύτερο σημείο κίνηση για την νομοθεσία ανεβήτρου έχουμε και καλύτερο σημείο κίνηση από ότι σε σχέση με αυτή την νομοθεσία που απασχολεί εμένα για τον τελικό εξοπλισμό. Θέλω να πω κάτι αυτή εξ αρχή πριν πω σε λεπτομέρειε τι αλλαγέ που προτείνω. Όχι καινοτομία μόνο για την καινοτομία, Θέλω γρήγορη πρόσβαση για τους ασθενείς, αλλά θέλω και ασφάλεια του ασθενούς. Και επισημαίνω ότι είναι θέλω γρήγορη πρόσβαση του ασθενούς, γιατί κάποιες εταιρείε παραπλανούν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τα μέλη του Κοινοβουλίου, προσποιούμενοι ότι ε, ουσιαστικά α, δημιουργείται πρόβλημα την πρόσβαση στην αγορά. Είναι ψέμα αυτό που λένε. Θέλουμε γρήγορη πρόσβαση στην αγορά Καθώς αυτό είναι πολύ σημαντικό, θέλω επίσης ε, ο τρικός θα πρέπει πρώτα να έχουν χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα, σε, πραγματική, σε πραγματικό στον οργανισμό και να έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι οι δισαγωγές. Προτείνω λοιπόν στην έκθεσή μου κάποιες σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν και θα αναφερθώ στις κύριες αλλαγές που προτείνω, ακριβώς για να χρησιμοποιήσω καλύτερα το χρόνο που μου δώσατε, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογή και η ταξινόμηση των συσκευών. Τροπολογίες 5, 22 και 140 για να μην υπάρχει γενική, γενικός των βιολογικών, αποκλείω τον κανόνα 31, διότι είναι συσκευές μοναδικές με διαλύματα άλλα τα μονολίπετα έπειτα οι 67 ε, και 79. Αυτή τη στιγμή να πω ότι είναι πρώτο σύστημα κοινοποίηση που ισχύει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διάκριση ανάμεσα στι συσκευέ διαφορετικών κλάσεων και να δούμε διαφορετικά την πρόσβαση στην αγορά. Χρησιμοποιώντας ε, τις ε, δοκιμές στο εργαστήριο ε, και τα αποδεικτικά στοιχεία που μας δίνουν πριν, υπάρχει, πριν μπουν στην αγορά. Τούτου λεχθέντος, εγώ προτείνω ένα σύστημα όπου σε κάποιες τομείς να χρησιμοποιεί συγκεντρωτική και αποκεντρωμένη δικαστή τα προϊόντα περιορισμένων επιδιαφορμής και μόνο τρει ε, συσκευέ και που μπορούν να φυτευτούν. Και αυτές ε, εξετάζω. Και έπειτα στην κλάση 2β και κλάση 3, δηλαδή προϊόντα υψηλού κινδύνου ή προϊόντα που εμφυτεύονται. Στην, στο 41α προτείνω κεντρική διαδικασία για η ιατρική υπηρεσία στο Λονδίνο να περιορίζεται, που περιορίζεται σε πολύ καινοτόμε εμφυτευτικέ ε, συσκευέ ή συσκευέ που συνδυάζονται με ιατρική ουσία. Και προτείνω και για τι μη καινοτόμε ε, συσκευέ την ίδια διαδικασία. Τρία λοιπόν μάλλον σύστημα τριών ε, ταχυτήτων, απλή κοινοποίηση πρώτα απ' όλα, δεύτερο σύστημα, αποκεντρωμένο και ε, κεντρικό σύστημα. Αυτό ως προσφορά από πλευρά μου, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω πραγματικά ότι το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει. Αν είσαστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τη δική μου γραμμή, και μπορούμε να βρούμε, αν θέλετε, και ένα συμβασμό κάπου μεταξύ μα, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και μια διαφορά σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά από ό,τι ισχύει σήμερα. Πάμε τώρα στι αρμοδιότητε ε, του φορέα κοινοποίηση. Κάποιοι βεβαίω ε, θα μου αντιτείνουν ότι αυτό που προτείνω εγώ θα οδηγήσει σε καθυστερήσει. Μα ήδη για την έγκριση των ιατρικών συσκευών σήμερα υπάρχουν μεγάλε καθυστερήσει. Η πρότασή μου προβλέπει για την ε, συγκεντρωτική διαδικασία κάτω από 9 μήνες διαδικασία για να μπει κάτι στην αγορά. Μια εικόνα για να δείτε τι ισχύει σήμερα. Ακριβώς για να διαψεύσω αυτά τα ψεύδη που έχουν δημοσιευθεί με πολύ προκλητικό τρόπο δηλαδή μπορεί ασθενή να περιμένει έω και τρία έτη, το οποίο είναι πραγματικά ανεύθυνο από, ιατρικές, από φαρμακευτικές κεντρικέ εταιρείε και από εσωτερικού κύκλου, γιατί αυτοί προέρχονται από κάποια λόμπι τα οποία πραγματικά πεχθάνομαι. είναι πραγματικά παραπλανών και ακολουθούν τι τακτικέ. Να σα δώσω λοιπόν μια ιδέα τι συμβαίνει σήμερα με τη βάση την κείμενη νομοθεσία, με βάση τη μελέτη για τη Κομισιόν και σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουν δώσει οι φορεί κοινοποίηση και οι εταιρείε, το σύστημα σήμερα χρειάζεται 2,5 με 4 μήνε κατά μέσο όρο για την κλάση 3 η νέα πρόταση της Κομισιόν προσθέτει σε αυτό το σύστημα όσο έχει αυτή τη στιγμή άλλους τρεις μήνες. Με τη διαδικασία ελέγχου κτλ. ώστε θα καταλήγουμε περίπου στους 7 με 8 μήνες. Η πρόταση δική μου προβλέπει έγκριση στην αγορά για την αποκεντρωτική διαδικασία 7,5 μήνες μέγιστο και για την αποκεντρωτική διαδικασία 9 μήνες μέγιστο. Άρα λοιπόν, ο ίδιος χρόνος για την κεντρική διαδικασία και δυόμισι μήνες παραπάνω για την κεντρική διαδικασία. Όποιος άλλος λέει κάτι διαφορετικό ψεύδεται. Εκτός βέβαια οποιοδήποτε είναι αφελής και δεν μπορεί να διαβάσει τα στοιχεία. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι εταιρείε να δείχνουν την ελάχιστη κοινωνική ευθύνη των ασθενών. Τώρα, πρόσβαση στην αγορά. Το επόμενο θέμα μα απασχολεί είναι ποιο δικαιούται να μιλάει για αυτό το θέμα και να σου λέμε αυτό. Φορεί τροπολογία Τροπολογίε 43-66 και 136-139. Ε, ό,τι και να συμφωνήσουμε αργότερα για την πρόσβαση στην αγορά αυτών των προϊόντων, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουν την αρμοδιότητα οι φορεί που δουλεύουν στον τομέα τη προ την αγορά. Αυτό είναι ουσιώδε. Δεν μπορεί ένα φούρνο να κάνει κοινοποίηση για, να για συσκευή για ένα γοπφό ή κάποιο που είναι υπεύθυνο ε, για την ασφάλεια του αυτοκίνητου σα να κάνει και την κοινοποίηση για ε, νιατρική σκευή. Περιμένετε, ε, είστε σίγουροι ότι ο οποίο σας με αυτά τα πράγματα έχει ειδική εμπειρία. Οπότε οι φορεί κοινοποίηση θα πρέπει να έχουν μονίμως προσωπικό, αρμόδιο ε, και εξειδικευμένο in-house και να έχει έχουν ειδικέ γνώσεις πάνω στον τομέα. Συχνά σήμερα κάνουν ανάθεση έργου εξωτερικά, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους αναθέτουν το έργο αυτό. Ε, αυτό λοιπόν, αυτός πρακτική θα πρέπει να περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό και οι κατάλογοι των ε, αναδόχων έρχονται να δημοσιεύονται. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο υπεργολάβος σε κάθε περίπτωση. Ο φορέας κοινοποίησης σε μια άλλη χώρα μέλος θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι είναι καταγεγραμμένος στα ε, αρμόδια εθνικά μητρώα. Και θέλω Είμαι σίγουρη και ότι οι προμήθειες και τα τέλη που ε, χρεώνονται να μας δίνουν συγκρίσιμα στοιχεία. Άρα πρέπει να κοινοποιούνται. Σήμερα μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση για εμφύτευση κοφού για 1.000 ευρώ σε μισή μέρα και να πληρώσει και 50.000 ευρώ και να περιμένεις 9 μήνες. Υπάρχει τέτοιο τεράστιο χάσμα. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Αυτή όμω είναι πραγματικότητα. Δεν κατεβάζω το κεφάλι μου αυτά που λέω. Έχω αποδείξει. Και το ξέρετε γιατί έχουν δημοσιευθεί και τέτοια παραδείγματα. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να αυξήσουμε, να, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των φορέων κοινοποίηση με το σύστημα που προτείνω, αλλά και σε οποιοδήποτε σύστημα τελικά σχέση. Ο φορέα κοινοποίηση είναι υπεύθυνο για τι ιατρικέ συσκευέ να έχει την κατάλληλη α, ιατρική δεξιότητα και την κατάλληλη φαρμακευτική δεξιότητα προκειμένου. Και τέλο, η επισήμανση, η καταθεσία των φαρμάκων που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και η επεξεργασία του. Σήμερα μιλάμε για απλή και πολλαπλή χρήση. απλή χρήση τι σημαίνει ότι μια συσκευή χρησιμοποιείται σε έναν ασθενή για μία και μόνο θεραπεία. Για μία αγωγή μάλλον. Και τέλος, αυτά τα προϊόντα απλής χρήσης είναι πολύ ακριβά και γι' αυτό συχνά επαναχρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχει όμως σαφές πλαίσιο και αυστηρό πλαίσιο σχετικά με την ε, επαναξεργασία και επαναχρήση τους. Και ποιος το κάνει αυτό. Η Κομισιόν κατεμέ δεν έχει μια σωστή ε, ταξινόμηση αυτών των συσκευών για απλή και πολλαπλή χρήση και δεν δίνει και τα κατάλληλα πρότυπα εν προκειμένου. Εγώ προτείνω συγκεκριμένε διατάξει. Για παράδειγμα, να είμαστε σίγουροι ότι μόνο οι συσκευέ που φέρουν την ετικέτα επαναχρησιμοποιούμενε θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πάλι. ώστε όλε οι συσκευέ κατά κανόνα να φέρουν την ετικέτα επαναχρησιμοποιούμενη και μόνο ο κατασκευαστή να μπορεί να βάλει την ετικέτα απλή και μόνη χρήση αν μπορεί να αποδείξει με βάση επιστημονικά πορίσματα γιατί αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Και να υπάρχει δυνατότητα ε, εταιρείε και νοσοκομεία πολύ συχνά να μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτόν τον ορισμό απλής χρήσης που έχει δώσει ο κατασκευαστής και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την ίδια συσκευή μετά από την επεξεργασία με απόλυτη ασφάλεια. Θέλω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να πω ότι οι συσκευές μονής χρήσεως χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά όταν δεν μπορούν να ε, τύχουν νέα επεξεργασία. Ιδάλω όλε οι συσκευέ να μπορούν να επεξεργαστούν με βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Αυτά είναι τα κύρια σημεία για την ε, κλινική έρευνα τώρα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στην τροπολογίες 25-59 και 89-96 με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα και το όφελο ασθενού που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν την Κομισιόν. Και θα πρέπει να υπάρχει έγκριση των κλινικών δοκιμών από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Βλέπετε και τις σχετικές τροπολογίες που σκόνουν και τις κλινικές δοκιμές. 97 και 102 οι τροπολογίες για την παρακολούθηση. Θέλουμε ένα σύστημα που να περιλαμβάνει ημερομηνία και τόπο ε, του περιστατικού. Αυτό ζητά ο ιατρικός κόσμος ε, γιατί μπορεί να υπάρχει ελάττωμα στην συσκευή, αλλά μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα να έχει υπάρξει σφάλμα από τον ε, αρμόδιο υπάλληλο. Ξέρω ότι ήμουν πάρα πολύ γρήγορη, ε, πρόεδρε. Πάντως δεν ακρηγόρησα. Βλέπετε ότι ζητούμε Πολλέ αλλαγέ στο κείμενο, τροπολογίες 1 ως 10 και τροπολογίες 100 με 119, ώστε το κείμενο να έρθει πιο κοντά στι δικέ μου απόψει. Με χαρά να ακούσω τώρα τι απόψει των συναδέλφων και των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπέρεντ, αρχίζουμε τώρα την παρουσίαση των συνεισηγητών. Η κυρία Μερή Μακίνε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την ξεκάθαρη τοποθέτησή της. Πρωτού σχολιάσω τις τροπολογίες, θα ήθελα να πω ότι ε, υπάρχει μια αναφορά στον Φεβρουάριο του 2012, όπου ο τότε ο Επίτροπος ε, σχεδίασε ένα σχέδιο δράσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Χρειάζεται αυτό να θεώρηση, διότι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε κάποια νεότερα αποτελέσματα για το τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη έχουν, ε, τους έχει ζητηθεί να κοινοποιήσουν την προέλευση των προϊόντων και να κοινοποιήσουν επίσης αξιολογήσεις που έχουν κάνει από ομάδες εμπειρογνωμόνων. Έχουμε κάποιες ενδείξεις σχετικά με το τι έχει συμβεί, με τις ε, επιτόπου επιθεωρήσεις, τις απροειδοποίητες. Έχουμε κάποια νεότερα για τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την ε, βελτίωση του συστήματος επαγρύπνησης που είχε ζητηθεί ε, και τις ε, πληροφορίες για τις παρενέργειες. Έχουμε κάποιες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες στον κλάδο αυτό. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει εξελίξεις, όμως θα ήθελα να μάθω τι κάνει η Κομισιόν για την παρακολούθηση του συστήματος, διότι όλοι ελπίζουμε σε μια βελτίωσή του, όλοι εργαζόμαστε για τον ίδιο στόχο, να βελτιώσουμε την ασφάλεια των ασθενών να θέσουμε σε κυκλοφορία στην αγορά τα καινοτόμα ε, ιατροτεχνολογικά προϊόντα για να είναι οι ασθενείς πιο ασφαλείς. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι ξεκάθαροι στόχοι, όμως ο καθένας ακολουθεί διαφορετικό δρόμο για την επίτευξή τους. Πρόεδρε, τώρα φτάνω σε ορισμένε από τι ιδέε που έχει υποβάλει η συγγήτρια. Την ε, προηγούμενη φορά ήμουν αρκετά προσεκτική και είπα ότι περιμένω ακόμα να με πείσουν για την, ε, συγκε... για την συγκεντρωτική ε, έγκριση. Καταλαβαίνω τη θέση της εισηγήτριας, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι οι τροπολογίες αυτές θα βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Θεωρώ ότι αν ενισχύσουμε εξίσου τις ε, αρμόδιες αρχές και τις αρχές εκκοινοποίησης, θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Και πιστεύω πως πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα στις αρμόδιες αρχές και στο τι εκείνες πρέπει να κάνουν και στο τι δεν κάνουν. Και να επίσης συγκεντρωθούμε στις, ε, στους εμπειρογνώμονες που έχουν αυτές οι αρχές ή που ενδεχομένως δεν έχουν. Πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, ρύθμιση και την βελτίωση του κλάδου. Τώρα όσον αφορά τις αρχές κοινοποίησης. Με ανησυχεί λίγο το σκεπτικό των ε, εμπειρογνωμόνων, των επιτοπίων εμπειρογνωμόνων σε αντιδιαστολή με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Γνωρίζω ότι πολλές φορές χρειάζεται κινητικότητα στην εμπειρογνωμοσύνη και ανανέωση των δεξιοτήτων. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν αυτό θα επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σίγουρα χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες στις αρχές αυτές. Αλλά πρέπει να προσέξουμε αυτοί οι εμπειρογνώμονες να συνεχίζουν να επιμορφώνονται. Τώρα, όσον αφορά τα τέλη, υπάρχουν δύο ειδών τέλη. Τα τέλη που ε, γνωστοποιούν κοινοποιημένοι οργανισμοί στις, ε, στις ε, επιχειρήσεις αυτές για τις υπηρεσίες τους. Και πραγματικά εδώ θα ήταν πολύ λυπηρό εάν παρατηρούσαμε το φαινόμενο του να κοιτάζουν την χαμηλότερη τιμή και να ψωνίζουν αλλά και επίσης να προσέξουμε να μην αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εδώ στην έκθεση. Τώρα όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης που είναι και το κύριο σημείο της πρότασης της εισηγήτριας. Κατά τη γνώμη μου περιπλέκει το σύστημα και δεν μας δίνει απολύτως καμία σαφήνεια και καμία εγγύηση για βελτίωσή του. Θα πρότεινα λοιπόν στις ε, τροπολογίες μου να κοιτάξω για το πώς θα ενισχυθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, επιθυμητό για όλους εξάλλου. Επίσης η εποπτεία μετά τη θέση σε κυκλοφορία στην αγορά είναι σημαντική. Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση των κοινοποιημένων οργανισμών και να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται με την νομοθεσία, ποια εφαρμόζεται και ποια τμήματα δεν εφαρμόζονται. Και πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι αυτό που υπάρχει εφαρμόζεται και κιόλα. Και θα ήθελα και γι' αυτό πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τη μία χρήση, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί εδώ. Διάβασα διεξοδικά την πρόταση της εισηγήτριας και Α το δω τώρα από την σκοπιά του ασθενή. Όταν μια εταιρεία διοχετεύει στην αγορά ένα προϊόν για μία και μόνο χρήση και εγώ βρίσκομαι σε, μια, σε ένα νοσοκομείο και βλέπω το νοσοκομείο να το πλένει και να το ξαναχρησιμοποιεί, αυτό θα με ανησυχούσε. Δηλαδή το σκεπτικό του όλα μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε μέχρι αποδείξεις του εναντίου μπορεί να είναι λογικό στη θεωρία, όμως δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και από πλευράς του παρασκευαστή και από ε, πλευράς του συστήματος ε, παροχής υπηρεσιών υγείας. Αναρωτιέμαι πραγματικά εάν οι ασθενείς, οι ομάδες ασθενών ε, έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δω κάποιες άλλες προτάσεις για αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά την σειρά του κειμένου δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα, μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό. Συνοψίζοντας πρόεδρε γιατί σας βλέπω με το σφυράκι στο χέρι, Βλέπω τους στόχους. Έχουμε κάποιες διαφορές ως προς το πώς θα τους επιτύχουμε και θα ακούσουμε και τα σχόλια των άλλων εισηγητών και πιστεύω πως θα βρούμε ε, συμβαστική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, Χόλγκερ Κράμερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισηγήτρια έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, μια εξαίρετη έκθεση, μια πολύ καλή βάση εργασία που μα οδηγεί προ τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να δώσει ε, πεδίο για συμβασμού στα σημαντικά καθοριστικά στοιχεία. Θα συμφωνήσω με την πολιτική σας ότι μπορώ να δεχθώ και εγώ όλε τι ε, κύριε γραμμέ τη εκθέσεω. Με τα τρία λεπτά που έχω στη μου, βέβαια δεν μπορώ να επισέλθω σε κάθε λεπτομέρεια, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα ασφαλώ. Θα ήθελα όμω να επισημάνω τη συνταξινόμηση των προϊόντων. Η πρόταση, στην πρόταση επιτροπή υπάρχουν κάποιοι κανόνε οι οποίοι είναι ασαφείς και οδηγούν και σε προβλήματα προ την ασφάλεια δικαίου. Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια λοιπόν. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα, θα συμφωνούσα μάλλον με τη διαγραφή του 21, αλλά και του 19 άρθρου, που αναφέρεται ή μάλλον μπορεί να οδηγήσει σε μια ε, περιττή διαφοροποίηση στα νανοηλικά, στην ταξινόμησή τους δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι ε, έχουμε μια σωστή κατεύθυνση, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ενίσχυση των προϋποθέσεων, των απαιτήσεων σε ορισμένες θέσεις, ε, όπως προτείνει και η εισηγήτρια, και στην ανάγκη για ε, εξειδικευμένη πραγματογνωμοσύνη στην κοινοποίηση ορισμένων προϊόντων. Χρειάζεται μια ασφαλώς πιο αυστηρή επιτήρηση της αγοράς για τα προϊόντα αυτά, για να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες συνέπειες και η ε, απέτηση είναι να συλλέγονται περισσότερα στοιχεία και να διατηρούνται αυτά σε βάση δεδομένων στη διάθεση βέβαια των κρατών μελών. Ξέρετε επίσης ότι δεν είμαι φίλος των προτάσεων αυτών, δεν ευνοώ τις προτάσεις αυτές που μιλούν για μια κεντρική διάρθρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Το ανέφερε και η κυρία Μαγκίνες. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Ροτσβέρεντ, το εάν ο άξονας πρέπει να είναι το συμφέρον της ασφάλειας του ασθενούς. Υπάρχει μια μελέτη από τη Βοστόνη για την ανάκληση ανακλήσεις προϊόντων. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα για την αδειοδότηση των προϊόντων στις ΗΠΑ. Αφορά λοιπόν τις ΗΠΑ η έκθεση αυτή, η μελέτη αυτή, συγκριτικά με, με την αγορά των, ε, την ευρωπαϊκή και δεν διαπιστώνεται διαφορά ως προς τη συχνότητα ανάκλησης ιατρικών προϊόντων. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγο ε, κάποιων περιστατικών περισσότερων προϊόντων από τις στις αυτό νομίζω θα πρέπει να μας δώσει τροφία σκέψη. Μια συμβαστική ιδέα λοιπόν ως πρόταση θα μπορούσε να είναι ε, να ξανασκεφτούμε αυτή την ομάδα συντονισμού για τα προϊόντα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να δώσουμε αρμοδιότητες στην Επιτροπή Συντονισμού για συγκεκριμένα προϊόντα, γιατί αυτό και θα επιβάρυνε το έργο της και θα το επιβράδυνε. Αλλά ίσως είναι η ομάδα αυτή, μπορεί να αποτελέσει η ομάδα αυτή συντονισμού τον κατάλληλο ε, εταίρο προκειμένου να συγκεντρώνονται και να ε, επαληθεύονται οι άδειες από τις διάφορους φορείς και οργανισμούς ανά την Ευρώπη που χορηγούνται γιατί όπως είπα δεν μπορεί ένας, ένα τέτοιο όργανο μυστικό να κάνει τα πάντα, αλλά μπορεί να συγκεντρώνει το υλικό και την σκηνοποίηση. Για το θέμα τώρα τη μίας χρήση. Μπορώ να συμφωνήσω με την εισαγήτρια, πιστεύω, όταν λέει ότι δεν είναι λογικό να ανατρέπονται οι οδηγίες χρήσεως για τα προϊόντα μίας χρήσης, γιατί ό,τι είναι μίας χρήσης πρέπει να παραμένει μίας χρήσης από την άλλη στην πράξη το να χαρακτηρίζεται, το να σημαίνεται ένα προϊόν ως μίας χρήσης, δεν φέρνει πάντα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην, στο εξή φαινόμενο, γιατί στη χώρα μου έχουμε πιο πολλά προβλήματα σε σχέση με τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων παρά με αυτά της μίας χρήσης. Επομένως, ανεξαρτήτως των ε, λύσεων στις οποίες θα καταλήξουμε, το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι βεβαίως να μην επαναχρησιμοποιούνται, να μην ανακυκλώνονται τα προϊόντα μιας χρήσης, αλλά και να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά και αυτά τις πολλαπλής χρήσης, δηλαδή να είναι με ψηλότερη ασφάλεια για τον ασθενή. Πάντως μπορούμε να περιμένουμε λύσεις συμβαστικέ, οι διαφορές μεταξύ μας είναι η κεντρική ή αποκεντρωμένη διαχείριση των αδειών, ε, και τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κράμερ. Βλέπω ότι έχει περάσει νερό στα βλάκι μετά τα ελαφρά εμπορικά ε, οχήματα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ριβασί, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια, διότι προτείνει η κυρία Ροτ Πέρεντ μία βελτίωση του συστήματος ε, σεβόμενοι πάλι τις ε, προθεσμίες που είναι πολύ σημαντικές για την διάθεση στην αγορά. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στη διαφάνεια της πληροφορίας, τον έλεγχο και την ε, διακυβέρνηση που είναι τα τρία σημαντικά για μένα θέματα. Για την ε, διαφάνεια καταρχάς κυρία εισηγήτρια θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο όσον αφορά τις κλινικέ δοκιμές και ιδιαίτερως στη διαβίβαση των δεδομένων για διεξαρτήσεις ε, κλινικές δοκιμές. Ε, όπως και στην οδηγία για τις κλινικές δοκιμές, εφαρμοστέως είναι ο κανονισμός 1049, δηλαδή το ύψιστο προϊό, ε, ο ύψιστος στόχος της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. Επίση, όταν θα μιλήσουμε για οργανισμού πιστοποίηση και αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν τα δεδομένα του και όχι σε συνοπτική μονομορφή. Εάν θέλουμε να μπορούμε να ελέγχουμε αυτού του οργανισμού πιστοποίηση, το στόχο αυτό τον επιδιώκουμε, τον ε, εξυπηρετούμε και χάρη στι μελέτε που δημοσιεύουν αυτοί, ε, ενώ συνήθω δεν τι δημοσιεύουν και δεν έχουμε πρόσβαση στι πληροφορίες αυτέ. Έλεγχη λοιπόν. Πώ θα γίνεται ο έλεγχο όλων αυτών των οργανισμών πιστοποίηση. Λέγεται ω λύση ότι θα τον αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Όμω, εγώ έχω πολλέ επιφυλάξει προ τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ενό κράτου μέλου και του οικίου οργανισμού πιστοποίηση. Και γι' αυτό έχω συστήσει μάλιστα με πολλούς επιθεωρητές, ε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η λύση είναι όταν υπάρχει μια προειδοποίηση ή ε, ένα συναγερμός σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να γίνεται η επιβεβαίωση, η επαλήθευση στον οργανισμό πιστοποίησης από τις αρχές του ειδικίου κράτους μέλους, αλλά και από το κράτος ε, το οποίο έχει γύρει το συναγερμό, πράγμα το οποίο μας δίνει μια, ένα διπλό, μια διπλή δυνατότητα ελέγχου. Επίσης, ε, με την ενημέρωση είτε από τους επαγγελματίες της υγείας, είτε από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, και πέρα από τις βιουταμέντ γιατί βεβαίως θα υπάρχει η ε, επαγρύπνησης προς τα φάρμακα, αλλά δεν είναι ο ασθενής εκείνος ο οποίος το συνηθέστερο θα δώσει τις πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω λέγοντας ε, για την διακυβέρνηση το συντονιστικό αυτό όργανο, ΣΟΙΠ, που απαρτίζεται από τα 27, των κρατών μελών κτλ. Ε, είναι μια πολύ ρευστή δομή. Δεν βλέπουμε ακριβώς ε, σε ποιο, ε, σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται. Αν κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά τι ΗΠΑ και το FDA, έχουν ένα διατακτικό που αφορά την ασφάλεια των φαρμάκων, αλλά και ε, κανονισμού ιατρική φύσεω. Και λέει η κυρία Ροτβέραντο ότι θα πρέπει να υπάρξει επαγρύπνηση προ τη διάθεση στην αγορά για την κατηγορία 3, αυτό την υποστηρίζω βεβαίω. Μα μιλάει για την κατηγορία 3, καινοτόμο κατηγορία 3 η κυρία Ροτβέραντο, θα πρέπει βέβαια αυτό να οριστεί. Αλλά όλοι οι εμφυτευόμενοι ε, και θεραπευτικοί ε, μηχανισμοί, το υλικό, το εμφυτευόμενο και ε, παρεμβατικό, ακόμη και αισθητικής φύσεως, ακόμη και καλλιντικής φύσεως και βλέπουμε πόσα προβλήματα έχουν προκύψει στον τομέα αυτών στη Γαλλία. Άρα λοιπόν, με μια κεντρική δομή που θα είναι αυτός ο ΣΟΕΠ, τα χασά που είμαι, θα υπάρχουν παράλληλα οι λύσεις ιατρικές οι οποίες καλύπτουν τόσο το, ιατρικό, ε, τόσο το φάρμακο όσο το ιατρικό προϊόν. Αλλά δεν είμαστε μέσα στην κατηγορία 3, την καινοτόμο, η οποία πρέπει να οριστεί ακόμη. Αποκεντρωμένα βεβαίως όλα αυτά. Κατηγορία 1, 2, 2α, καμιά αντίρρηση, ας είναι αποκεντρωμένα. Αλλά όταν έρχεται κάποιος να εμφυτεύσει ένα ιατρικό ε, μηχάνημα ή εξοπλισμό στο σώμα σας, ε, κάποιος θα πρέπει να το παρακολουθεί αυτό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε σε μια γκρίζα ε, ζώνη. Επίσης, για αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι καρκινογόνα, διαταρακτές ενδοκρινολογικοί, μεταλλακτικά και όλα αυτά θα πρέπει ιδιαίτερα να τα χειριστούμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε δηλαδή, στη γενική κατηγορία. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της κυρίας Γιανακουδάκη, θα ο κύριος Τσάρμανο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να στήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου μου που δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Θα μιλήσω εξ ονοματός του για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Εμείς συζητούμε εδώ ε, αυτά τα προϊόντα μαζί με τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα αλλά όμως πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο. Διαφορές οι οποίες ε, πρέπει να τις δούμε, πρέπει να και πρέπει να ρυθμιστούν. Πιστεύω ότι ένας κανονισμός θα μας, θα μας έδινε μεγαλύτερες δυνατότητες για, να, για διορθωτικά μέτρα. Καταρχάς η ποιότητα της αγωγής και η ασφάλεια των ασθενών είναι υψίστες προτεραιότητες. Από την άλλη όμως πρέπει να φροντίσουμε και για το σύστημα υγεία και την διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών στο σύστημα αυτό. Χρειάζεται να υποστηρίξουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, με καλύτερη ποιότητα και την επαρκή διάθεση των προϊόντων αυτών. Και να μην εμποδίσουμε λοιπόν τις ε, υπηρεσίες υγείας με υπερβολικές ρυθμίσεις. Πιστεύω ότι η πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα, δεν θα μας οδηγήσει σε μια αποδοτική και σωστή δομή. Θα αυξήσει την γραφειοκρατία και έχουμε ήδη ορισμένα εργαλεία. Για παράδειγμα, τις ε, ε, τους κοινοποιημένους οργανισμούς ε, και τις επιστοποίησεις συμμόρφωσης. Και πραγματικά δεν θα πρέπει να είμαστε αντιπαραγωγικοί. Χρειαζόμαστε ικανούς οργανισμούς, αρμόδιους οργανισμούς, τους οποίους θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Εάν όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου, τότε πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος από αυτούς ε, τους ε, αρμόδιους θα είναι εκείνο που θα τα ελέγξει. Τώρα, όσον αφορά τις, ε, την ταξινόμηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για παράδειγμα, μηχανήματα για την, για την μέτρηση της πίεσης. Αυτά είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούν, για παράδειγμα, να συνδεθούν με ένα τηλέφωνο για την μετάδοση των δεδομένων. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν αυτό το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό ή όχι. Και να δούμε τι γίνεται τώρα και με το λογισμικό. Είναι το λογισμικό απαραίτητο συστατικό ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή όχι. Εγώ είμαι γιατρός. Και εδώ και εννέα χρόνια δουλεύω στην ε, μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όσον αφορά τα μίας χρήσης προϊόντα, έχω, έχω κάποια εμπειρία από αυτό. Και τι μας λέει λοιπόν η πρακτική τους εφαρμογή. Πιστεύω πως πραγματικά οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές πρέπει να είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν αν αυτά τα προϊόντα θα είναι μίας χρήσης ή όχι. Ε, πιστεύω πως είναι καλύτερο αυτή η επανεπεξεργασία να λάβει χώρα. Έχω δει πολλές φορές, για παράδειγμα, καθετήρες ή διάφορα, διάφοροι να πλένονται από τις ε, νοσοκόμες το βράδυ και να ξαναχρησιμοποιούνται. Και πραγματικά σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν είχαν άλλη επιλογή, δεν υπήρχαν άλλα προϊόντα στη διάθεσή τους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ και να χαιρετήσω την αγαπητή συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε για αυτό το θέμα. Είναι πολύ δύσκολο και περίπλοκο αυτό το θέμα, αλλά ήταν πραγματικά αναγκαίο σε αυτό το τομέα να αναθεωρηθεί η φυστάμενη νομοθεσία. Και είναι πολύ λογικό σαν το γεγονό ότι ουσιαστικά ξαναγράψατε από την αρχή, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό την πρόταση τη Επιτροπή και το κάνετε με πολύ λογικό ε, τρόπο. Πιστεύω ότι η διαδικασία που έχουμε ενώπιόν μας για συζήτηση επί του θέματος θα μας επιτρέψει να μπούμε στις λεπτομέρειες διαφόρων πτυχών της πρότασης. Εγώ θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ επίσης για όσα είπατε για την έγκριση, για την πρόσβαση στην αγορά, τη διαδικασία που προτείνεται. Τα θέματα των κλινικών ερευνών και τις κλινικές δοκιμές όπως τις προτείνεται, που μπορεί να μας δώσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την χρησιμότητα και την ασφάλεια των ε, ιατρικών αυτών προϊόντων, Και όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και από μια συγκεκριμένη διοντολογία, κώδικα διοντολογίας. Τώρα το θέμα των φορέων κοινοποίηση είναι πραγματικά περίπλοκο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα υψηλού κινδύνου ή τα προϊόντα εκείνα που είναι, αν θέλετε, σε πειραματικό στάδιο είναι καινοτόμα, είναι πραγματικά λογικό η έγκριση να συνδέεται με έναν πιο συγκεντρωτικό φορέα κοινοποίηση. Και αυτό βεβαίω συνδέεται με την δομή που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και το σύστημα ε, εγκρίσεων που δίνουν και για άλλες κατηγορίες ε, για προϊόντων. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία που έχουμε από άλλα προϊόντα, όπως χημικά προϊόντα ή θα θυμάστε πρόσφατα, ε, την ε, έκθεση που υιοθετήσαμε για τις ενδεκρονολογικές ε, και σουσίες και συζητήσαμε και πάλι και εκεί τους κινδύνους που ελοχεύουν από, από τη χρήση τέτοιων ουσιών. Χρειάζεται λοιπόν να ε, υπογραμμίσουμε αν θέλετε ε, έντονα και με κόκκινο χρώμα αυτές τις συσκευέ καθώς ε, πραγματικά μπορεί να είναι υψηλού κινδύνου. Σε ό,τι αφορά τώρα πάλι την έγκριση τη διαδικασία έγκριση αυτών των προϊόντων. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με τα κριτήρια που επέλεξε η συγγήτρια, όμω θεωρώ ότι δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και κάποιες άλλες πτυχές που γύρουν ερωτηματικά. Γιατί δεν είναι οι ίδιοι οι ασθενείς που θα πάνε να εξετάσουν ε, την ετικέτα που φέρει ε, το προϊόν, αλλά οι γιατροί θα το κάνουν αυτό. Έχω δηλαδή κάποια ερωτηματικά σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε ειδικά για τις συσκευές μονής χρήσης. Αυτό ισχύει πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις και όχι να αποστέλλονται σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εκεί επαναχρησιμοποιούνται. Πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε μια πρώτη ύλη και μια πολύ καλή συζήτηση και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό, εξαιρετικό μάλλον τελικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, συνάδελφοι, περνάμε στον επόμενο κύκλο. Έχει ο καθένα δύο λεπτά στη διάθεσή του, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσει η Κομισιόν να πάρει και εκείνη το λόγο. Έχουμε και μετά την έκθεση του κυρίου Λίζα να συζητήσουμε, που κινείται στα ίδια πλαίσια. Καταρχά, έχει... πρώτη έχει το λόγο η κυρία Κούκοβιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. πραγματικά χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Και η εμπειρία μου δείχνει ότι το πρώτο πρόβλημα και το κυριότερο είναι η διαφάνεια. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαφάνεια στα κρατημέλη. Και πιστεύω ότι εξαιτίας αυτού πρέπει εμείς εδώ να δημιουργήσουμε ένα είδος ενιαίας εσωτερικής αγοράς, διότι συζητούμε για άλλες ε, πτυχές της εσωτερικής αγοράς, αλλά όχι για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι μια πρόκληση τα προϊόντα αυτά για εμάς. Και βέβαια το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά. Με μια κεντρική έγκριση, το ερώτημα που έχω εγώ είναι το πόσο χρόνος θα χρειαστεί για την όλη διαδικασία, διότι πάντα, τα πάντα είναι ζήτημα χρόνου. Πότε δηλαδή θα μπορεί ο ασθενής πόσο γρήγορα να έχει αυτά τα προϊόντα στη διάθεσή του. Και επίσης, πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες. Και τέλος το ζήτημα της ε, πραγματική ε, εφαρμογής, τη εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο, υπό κανονικές συνθήκες, τι γίνεται εκεί. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε βελτιώσεις, χρειαζόμαστε κάποιο, κάποιο είδους μπούσουλα, αν θέλετε, αλλά δεν ξέρω εάν η κεντρική αδειοδότηση είναι η κατάλληλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Πανάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Γιατί μέλημά της είναι πάνω απ' όλα η ασφάλεια του ασθενούς, μια προσέγγιση που επικροτώ και εγώ. για την αποκεντρωμένη αξιολόγηση πριν από τη διάθεση στην αγορά. Για να αποφύγουμε τον κατακλυσμό μιας κεντροποιημένης διαδικασίας από μέτρητα προϊόντα θα πρέπει νομίζω να αναφέρουμε, να ορίσουμε κριτήρια της κατηγορίας 3 συν και να αναφέρουμε τα ε, προϊόντα εκείνα, τα ιατροτεχνολογικά της κατηγορίας 3 που δεν θα χρειάζεται να υπαχθούν στην ε, κεντροποιημένη διαδικασία. Επίσης, οι μηχανισμοί πιστοποίησης δυστυχώς δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό και ικανότητα να παρακολουθήσουν τις τεχνικές απαιτήσει των νέων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τις στηρίσουν. Δεν έχουν επαρκή εμπειρία για την επαλήθευση της ποιότητας των κλινικών ε, ε, εξελίξεων και ίσως χρειαστεί να απευθυνθούν σε εξωτερικές αναθέσεις. Το παράδειγμα της FDA των ΗΠΑ έχει αναφερθεί αρκετές φορές. Θα ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν έχει αδειοδοτηθεί και εγκριθεί από την FDA και στη συνέχεια απεσύρθησαν από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω σοβαρών προβλημάτων. Επίσης η FDA έχει εντολή να προστατεύει και να προάγει την δημόσια υγεία ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν ε, ενώ οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν τον ίδιο, το, το ίδιο καθήκον. Για δε η συντονιστική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ε, καθοριστική γνώμη, δεν έχει αποφασιστική ε, αρμοδιότητα και όσο δεν μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα ή τους κινδύνους. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποια κριτήρια για την κατηγορία 3, μια δεύτερη κατηγορία 3 που θα αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και ε, ιατρικά και ιατροτεχνολογικά. Επίσης θα χρειαστεί μια εξειδικευμένη σήμανση στη μία χρήση, γιατί η σήμανση στη μία χρήση μπορεί να οδηγεί σε παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και πιστεύω ότι θα χρειαστεί ίσω κάποια στιγμή να μα απασχολήσει ένα χωριστό νομοθέτημα. Εν πάση περιπτώσει όμω, για να μην, να μην παίζουμε με την ασφάλεια. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο, ο πρόεδρο, ο επόμενο ομιλητή. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Η συζήτηση διαξάγεται σε χρονική στιγμή όπου στη Γαλλία έχει ξεκινήσει η δίκη του Ζων Κλωτμάς, του ιδρυτή της εταιρείας PIP, στην οποία απευθύνθηκαν πολλές γυναίκες και αυτές είναι στο μυαλό μου όσο σας μιλάω, ο κύριος Πίπνο μόνος ο οποίος βρίσκεται στο εδόλιο γιατί κανείς άλλος συγκατηγορούμενος του δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν είχε αρνηθεί η αρμόδια υπηρεσία την πιστοποίηση ε, αλλά στη συνέχεια το 2005 δόθηκε η πιστοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθησε η Γαλλία το 2007. Με το κείμενο λοιπόν που έχουμε στη θέσή μας μπορεί να κινδυνέψουμε να δούμε μια νέα υπόθεση ΠΙΠ. Η φιλοσοφία του ρύθμιση στηρίζεται στην ευθύνη του φορέα και μάλλον του πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, του εμπλεκόμενου φορέα και δεν έχουν οι δημόσιες αρχές, οι κρατικές αρχές δυνατότητα επέμβασης. Χωρίς όμως συντονισμό, χωρίς κυρώσεις, είναι μόνο πλασματική η δυνατότητα προστασίας. Ενώ βρισκόμαστε σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, με προσπάθεια για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εμένα πρέπει να τις βοηθήσουμε σε αυτό, αλλά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο πάνω απ' όλα την ασφάλεια, αλλά και την εμπιστοσύνη. Η υπόθεση PIP δείχνει ποια είναι τα προβλήματα ως προς την επιτήρηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς, η παραγωγή θα πρέπει κατά τρόπο απρόβλεπτο, απροειδοποίητο και τακτικό να ελέγχονται. Η ποιότητα παραγωγής θα πρέπει να εξετάζεται στη διαδικασία ελέγχου κατά την πιστοποίηση του προϊόντος και αυτό σημαίνει και την διάδοση των σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Κάθε αντίθετη πληροφορία θα πρέπει να παραμένει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ε, και η υπόθεση ΠΙΠ θα πρέπει να αποτελέσει ένα υγειονομικό ηλεκτροσόκ, κύριε Πρόεδρε, όταν έχουμε από το ε, British Medicine Journal αντίστοιχες αναφορές για προβλήματα που εμφανίζονται στην Τσεχία, νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει, όπως είπε ο κύριος Κράμερ, να αυτοματικοποιηθεί η ε, διάθεση των, σήμανση των προϊόντων μίας χρήσης. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα πολύ ολιστηρό πεδίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λίσσα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Ροτ Μπέρεντ για την δουλειά της και για τις ε, παρατηρήσεις εκ μέρους του ΕΛΚ τις οποίες συμμερίζομαι. Πιστεύω πως όλοι πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία και να προστατεύσουμε περισσότερα τους ασθενείς. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα με την κυρία Ροτ Πέρεντ και στις ε, εκθέσεις και τη δική της και τη δική μου υπάρχουν ε, αρκετές ε, όμοιες προτάσεις. Είμαστε σε σχεδόν παράλληλη γραμμή. Πιστεύω πως η αλλαγή της σειράς της έκθεσης είναι λογική, τη συμφωνώ μαζί της. Επίσης πιστεύω ότι η εμπειρογνωμοσύνη των κοινοποιημένων οργανισμών πρέπει να ενισχυθεί Τώρα, εάν θα ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη διατύπωση τη εισηγήτριας ή μια άλλη, ε, θα το δούμε. Αλλά πρέπει σίγουρα η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει πιο σαφή. Τώρα, όσον αφορά τις, ε, τον κανόνα τη μια χρήση, είμαι κάπω αμφίβολο γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρο. Καθώ επίση και αυτό που ανέφερε ο κύριο Κράμερ για τα νανοσωματίδια. Εδώ ε, είμαι κάπως σκεπτικός. Επίσης, συμμερίζομαι την άποψη της Μερή και κάποιων άλλων για την ε, μη ε, κεντρική αδειοδότηση Πιστεύω πως η καινοτομία στην Ευρώπη θα ε, δρομολογηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν σκάνδαλα, όντως, όχι μόνο από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και για φάρμακα. Να σας θυμίσω ότι έγινε με τα αντισυλληπτικά πριν από κάποια χρόνια και πραγματικά ε, είδαμε τι έγινε εκεί και θα μπορέσουμε να μάθουμε από αυτό. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για διαπραγμάτευση. Χρειαζόμαστε χρόνο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα τρία ε, χρόνια, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα αυτά μας στάσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σνέλαρτ. Κύριο Σνέλαρτ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσεις της ηγήτριας και αποδεκτέ στο μεγάλο του βαθμό. Θα επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία μόνο για την αναδιάρθρωση των κεφαλαίων, τη σειρά των κεφαλαίων καλύτερα ναι. Η αναδιάθεση, όταν έχουμε να κάνουμε με μία ε, σύγκρουση στην οποία ο παραγωγός μιλάει μόνο για μία χρήση και προσπαθεί να πουλήσει το προϊόν του και άρα μπορεί να έχει ένα αντικείμενο τη δυνατότητα να το ανοίξει μόνο μία φορά και μετά να μπορεί να ξανακλείσει, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή μόνο για μία φορά. Αυτό θα μπορούσε, εάν εξασφαλιστεί δυνατότητα για την ε, αξιοποίηση και επανάληψη τη χρήση, να μειώσει σημαντικό, σημαντικά το κόστο τη παραγωγή. Άρα, ίσω θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση με τα προϊόντα τα οποία έχουν περάσει από μια νέα επεξεργασία και είναι έτοιμα για δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα πρέπει, ε, αυτή η διαδικασία της αξιοποίησης, της ε, ε, αποκατάστασης να επαφεθεί μόνο στα νοσοκομεία ή αν θα πρέπει να επιστρέφει το προϊόν στον παραγωγό. Επίσης είμαι κάπως επιφυλακτικός για το αν η διαδικασία της πιστοποίησης της ε, άδειας, ε, της αδειοδότησης μπορεί να επαρκεί και να είναι ικανή για την διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων. Το σύστημα νομίζω όπως το προτείνεται μπορεί να λειτουργήσει αλλά στους ελέγχους θα ήθελα να είμαστε κάπως πιο αυστηροί να ορίσουμε τέτοια συστήματα με αδιασφαλιστικές δικλίδες, επί παραδείγματι απροειδοποίητους ελέγχους, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για να είναι και επαληθεύσιμο το αποτέλεσμα του ελέγχου, για να αποφύγουμε νέα ιατροφαρμακευτικά σκάνδαλα και να υπάρχει, όπως είπα, απροειδοποίητος δειγματοληπτικός έλεγχος. Αυτό είναι μια απαραίτητη προειδοποίηση, ε, προϋπόθεση. Και ίσως θα μπορούσε κάποια στιγμή να θεσπιστεί ένας εθνικός φορέας στην Ευρώπη, ο οποίος θα ελέγχει τους ελεγκτές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε έτσι τον κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Σφανούκ είναι η νέα διευθύντρια από, την μονάδα, από τη Διεύθυνση μάλλον, ε, Θεμάτων του Καταναλωτού. Την καλωσορίζουμε εδώ. Η κυρία Λετενιέ επίσης έπρεπε να ομιλήσει σε κάποια διεθνή διάσκεψη. Τώρα βλέπω όμως ότι είστε εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ. Μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα για αυτή τη συζήτηση να ακούσουμε τις απόψεις σας που είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και πρώτη φορά που είμαι παρούσα εδώ να σας πω ότι έχω μια σαφή πολιτική εντολή από το βρεστάμενό μου πράγματι και εμείς θέλαμε να κάνουμε μια παρακολουθήση της ε, αυτού του τομέα πολιτικής. Ήταν μείζονο σημασία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τι προτάσει που κάνατε. Και εμεί με το ίδιο σκεπτικό κάνουμε την πρότασή μα και με τα διδάγματα που αντλήσαμε, όχι μόνο με το σκάνδαλο του ΠΙΠ, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε ευγνώμονε γιατί ετέθη το ερώτημα τι κάνουμε, πού είμαστε με το σχέδιο δράση που προτείναμε πέρυσι, αλλά πρόεδρε αν μου επιτρέπετε να το αφήσω αυτό στο τέλος, αν έχω το χρόνο, ιδάλλως, ε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Επί των θεμάτων που ετέθησαν συζήτηση βεβαίω, η έγκριση για την αγορά είναι ένα θέμα και όλη η δουλειά που κάναμε στην πρότασή μας είχε πάντοτε υπόψη το εξή. Πώς θα βελτιώσουμε την ασφάλεια του ασθενούς με την όλη διαδικασία αδειοδότησης. Ήδη εδώ το έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, επί τη ευκαιρία των πολύ χρήσιμων εργαστηρίων που διοργάνωσε η συγγήτρια και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πόσο ε, σημαντικό είναι αυτό το θέμα και ποιο προσφύλλο πρέπει να το διέπηκε. Και μελέτη τύπου ε, είχαμε σαφή αποτελέσματα ότι ό,τι και αν προτείνουμε θα έχει σκοπό την αύξηση της ασφαλείας για τον ασθενή. Και το σύστημα έγκρισης δεν θα γίνει πιο χρονοβόρο ε, και λιγότερο ασφαλές για τον ασθενή. Άρα λοιπόν η ασφαλή του ασθενού είναι ε, το πρώτο και το μείζον. Δεν είναι μόνο η αγωνιστικότητα του κλάδου που και αυτό είναι σημαντικό βεβαίω, αλλά εκεί αποκλίνουμε ε, σημαντικά από την φιλοσοφία. Κατανοούμε βεβαίω την ευαισθησία τη ηγήτρια και όλα τα θέματα που θέτει, αλλά σε άλλα σημεία της πρότασης μπορούμε να ε, κάνουμε κάποιες αλλαγές για να αυξήσουμε τον πύχη σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της ε, προστασίας και της ασφάλειας. Και πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε με αυτόν τον τρόπο τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία των προϊόντων, κατανοούμε τι ανησυχίε που ακούστηκαν και πράγματι πολλά από αυτά που ακούστηκαν σήμερα είναι πολύ λογικά πράγματα. Αλλά όπως ήδη είπαν και πολλοί συναδελφοί σας, ε, υπάρχει και το θέμα της σκοπιμότητας. Αν θέλουμε να κάνουμε πολύ εξειδικευμένη τεκτοθεσία, θέλουμε να επιλέξουμε την ε, μονή ε, χρήση ή την πολλαπλή χρήση, θα πρέπει τελικά αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε να είναι εφικτό και εφαρμόσιμο. Για τον κανόνα 31, με χαρά να σας δώσουμε περαιτέρω εξηγήσει στόχος μας, δεν είναι προϊόντα ε, μηδενικά σε κίνδυνο. Μιλάμε για προϊόντα που σε συγκεκριμένες κατηγορίες που ορίζονται με απόλυτη ακρίβεια θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της ασφάλειας και γι' αυτό ταξινομούνται με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι αφορά τις ε, κλινικές έρευνες, ήδη ε, και εσείς εδώ είχατε πολλές συζητήσεις, τις παράλληλες συζητήσεις για τις κλινικές δοκιμές, για αυτό το με και με χαρά. Μπορούμε να πούμε, λαμβάνοντας υπόψη όσα λέγονται από την Επιτροπή Διοντολογίας, να λάβουμε υπόψη να όλα αυτά, επαναλαμβάνω, στην πρόταση για τι κλινικέ δοκιμέ, Ό,τι αφορά του φορεί κοινοποίηση, πράγματι, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι να λαμβάνουν αποφάσεις και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δίκιο έχετε σε ό,τι αφορά τα τέλη. Κατανοούμε τα σχόλια σα, πράγματι, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Το ίδιο για την επαγρύπνηση και εποπτεία τη αγορά. Και για μα είναι στοιχείο κλειδί για την εφαρμογή τη νομοθεσία και εδώ και πάλι ε, μπορούμε να δεχτούμε πολλά από όσα ε, προτείνατε, κινούνται προς την κατεύθυνση με τη δική μας πρόταση και με χαρά να προσαρμόσουμε το δασί μας και ώστε να αυξήσουμε το, ε, τα τα θέματα ενημέρωσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ό,τι αφορά την σειρά των κεφαλαίων. Εντάξει, η Επιτροπή σας θα αποφασίσει αν είναι πιο λογικό να είναι άλλη σειρά ε, στη δομή της πρότασης. Αυτό δεν αντίκειται στην ουσία ε, της πρότασης. Οποιοδήποτε λοιπόν ε, βελτίωση στη λογική της πρότασης με χαρά τη δεχτούμε. Τώρα τι έχει γίνει από πέρυσι. Θα γνωρίζετε. Και ίσως έτσι απαντώ και σε κάποια ερωτήματα που ακούστηκαν σήμερα. Όταν ε, ξέσπασε το σκάνδαλο γιατί πραγματικά ήταν ένα σκάνδαλο, ήταν καθαρή απάτη, κάναμε μία δοκιμή αντοχής, ένα stress test για να δούμε κατά πόσον η πρόταση που κάνουμε τώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ε, και να αποφύγουμε αν θέλετε αυτό το σκάνδαλο αν υπήρχε νομοθεσία τότε και το ε, η απάντηση ήταν θετική αυτή τη δοκιμή και γι' αυτό στην πρώτη μα ανακοίνωση, όταν προτείναμε αυτή την αναθρομοθεσία είπαμε ότι λάβουμε υπόψη το σκάνδαλο ΠΙΠ και ελπίζουμε ότι όταν θεθεί σε εφαρμογή αυτή νομοθεσία δεν θα ξανασπάσει το σκάνδαλο. Επίση, φέτο κάναμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις τις οποίες είχαμε υποσχεθεί. Ήδη έχουν γίνει κοινή ανεξάρτητη έλεγχη από την Κομισιόν με την Υπηρεσία Εκτινιατρικών που ε, προσέθεσε στην εντολή του τη δυνατότητα να κάνει σε εθνικό επίπεδο ανεξάρτητος ελέγχους. Τέσσερις χώρες έχουμε περάσει από ανεξάρτητο έλεγχο ήδη και θα προχωρήσουμε τους ελέγχους. Ό,τι αφορά την ίσχυση των κριτηρίων για τους φορείς κοινοποίησης, τα κριτήρια μάλλον που θα πρέπει να επαληθεύουν οι φορές και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι φορές σε λίγους μήνες πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να σας ανακοινώσουμε τα κριτήρια αυτά. Για να τελειώσω το χρόνο μου, λοιπόν. Ε, αυτή τη στιγμή εκπονούμε ένα έγγραφο, το οποίο ελπίζουμε να είναι έτοιμο έω το καλοκαίρι, το οποίο θα περιγράφει ό,τι έχουμε κάνει σε σχέση με το σχέδιο δράση, το οποίο δεν έχουμε ξεχάσει. Το δουλεύουμε παράλληλα με την πρόταση αυτή. Ε, με χαρά να έρθουμε και να σα το παρουσιάσουμε το σχέδιο δράση, αν το κρίνετε αναγκαίο. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι στο καλοκαίρι, αλλά 60-70% ε, του σχεδίου είναι έτοιμο και με χαρά είμαι σε διάθεσή και για άλλε ερωτήσει. Ευχαριστώ, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ντάκμαρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βέβαια δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα όσα υπόθηκαν αλλά θα επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα. Πρόσβαση στην αγορά, γιατί αυτό έθεσε αρκετά σαν αρκετοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή για άλλη μια φορά, το χρονοδιάγραμμα. Από την αξιολόγηση συνεπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι να μπει ένα προϊόν στην αγορά πέραμε τέσσερις μήνες. Με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προστίθενται ακόμη τρεις μήνες, δηλαδή συνολικά έχουμε επτά μήνες χρονοδιάγραμμα για να διατεθεί ένα προϊόν στην αγορά. Η δική μου πρόταση με πολύ συγκεκριμένες ημέρες, δίλε ημέρες, μετρήσιμε, λέει μια κεντροποιημένη διαδικασία. Για τις ε, διαδικασίες της Εθνικές Αρχές 7 μήνες την αποκεντρωμένη διαδικασία, διορθώνει η ομιλήτρια, και εννέα για την κεντρική διαδικασία. Επτά μήνες για την αποκεντρωμένη στις εθνικέ ε, αρχές και εννέα για την κεντρική. Άρα δεν υπάρχει καθυστέρηση προ τη διάθεση στην αγορά, δεν υπάρχει αμφιβολία ω προ αυτό. Όποιο ισχυριστεί ότι μπορεί να κρατήσει τρία χρόνια αυτή η διαδικασία, απλώ δεν λέγει την αλήθεια και δεν πρέπει να παραπλανούμε ούτε τους ε, ασθενείς, ούτε τις οργανώσει των καταναλωτών, ούτε και τους εαυτούς μας. Οποιοςδήποτε λοιπόν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι καλού τύπου και επίπεδου lobbying αυτά που ακούγονται. Επίσης κεντροποιημένος, αποκεντρωμένος, ένα ζήτημα, ένα δίλημα το οποίο είπε τώρα από το θέσατε και ο Αντώνιο και όλου ουσιαστικά, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στο δικό μου το έργο και βέβαια αναφέρομαι σε οτιδήποτε εμφυτεύεται που αναφέρει η κυρία Ρίβαζη, προϊόντα της κατηγορίας 3 δηλαδή, μιλάμε για το 20% του συνόλου των προϊόντων. Πολύ μικρό ποσοστό, 20% των προϊόντων που διατίθενται συνολικά στην αγορά για... και πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την ε, λεπτομέρεια. Ο κύριος Λίσε είναι αυτός ο οποίος ανέφερε τη δυνατότητα για μια συμπληρωματική κλάση 3, 3+, εγώ δεν έχω αντίρρηση ως προς την εξέταση των ορισμών αυτών, το πώς θα τους ορίσουμε, αλλά οτιδήποτε εμφυτεύεται και παραμένει εντός του ανθρωπίνου σώματος και συνδέεται με ένα ενεργό συστατικό, φαρμακολογική ουσία δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλεται σε μια διαδικασία αντίστοιχη και ισοδύναμη με αυτή των φαρμάκων γιατί παραμένει ενεργό μέσα στο σώμα, μέσα στον οργανισμό με μια ενεργή ουσία φαρμακευτική θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Είτε πρόκειται για την παρίνη που μπαίνει στο αίμα για να μα προστεύει από τη θρόμβωση, είτε για οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το προϊόν λειτουργεί σωστά και αυτή είναι ακριβώ η διάκριση στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Είτε πρόκειται για αποκεντρωμένη, είτε πρόκειται για κεντρική διαδικασία, είτε πρόκειται για εθνικέ αρχέ, είτε πρόκειται για Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, χρειάζεται και δεν είναι αυτό το ζήτημό μου το να υπάρχει μια διαφοροποιημένη διαδικασία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μπορώ να διακρίνω ανάμεσα στον ναρθικά, στον ε, γύψο και την ινσουλίνη είτε μπαίνει με την ε, ένεση στο σώμα είτε μπαίνει με το ε, εμφύτευμα. Αυτό είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Η διαδικασία, και αυτό θα το καταλάβει ο καθένα, η διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κατά βάθο εσφαλμένη, βαθύτατα εσφαλμένη. Οι οργανισμοί, οι διάφοροι, βεβαίω δεν έχω καμιά αντίρρηση, πρέπει να του αναβαθμίσουμε, δεν έχω καμιά αντίρρηση να του αναβαθμίσουμε. Αλλά εάν δεν επιμείνουμε να έχουμε εσωτερικέ πραγματογνωμοσύνε, πάντοτε θα εξαρτώμεθα από του υπεργολάβου. Και πώ θα ξέρουμε ότι είναι καλή, πώ θα ελέγχουμε, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου. Οι εθνικέ ε, αρχέ μπορεί να έχουν έλεγχο στι αρχέ κοινοποίηση, αλλά όχι στου υπεργολάβου του. Και έτσι έχουμε σαφέστατες δυνατότητες να επισέλθει, να παρισφρήσει σφάλμα και να φτάσουμε μέχρι την καταστροφή τι, τι ιδέα μπορεί να έχουμε για αυτούς τους υπεργολάβους και το, το, γνωστικό τους υλικό. Πώς μπορούμε να κοινοποιήσουμε, πώς τολμάμε να κοινοποιήσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει ελέγξει ένας γιατρός, ένας, ένας ε, φαρμακοποιός, ένας ειδικός της έρευνας πώς μπορούμε να αδειοδοτήσουμε, να ετοιμάσουμε την αδειοδότηση ενός προϊόντος εφητευωμένου στο σώμα όταν δεν έχουμε ιδέα για την ιατρική λειτουργία του προϊόντος αυτού και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιδράσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και είναι απαράδεκτο επίσης ο, οργανισμός αδειοδότησης να είναι μόνο μία ομπρέλα πίσω από την, κάτω από την οποία κρύβονται πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης, πολλοί από εσάς αγαπητοί συνάδελφοι αναφερθήκατε στους ελέγχους και την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην χώρα. Ναι, αλλά ποιο το κάνει αυτό. Αυτό το κάνουν οι εθνικέ αρχέ, το κράτο. Και ποιο το πληρώνει, όλοι μα. Όλοι πληρώνουμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι περιττό εάν η αδειοδότηση και η πρόσβαση στην αγορά γινόταν με σωστού κανόνε. εάν υπήρχε σωστός έλεγχο πριν από την πρόσβαση στην αγορά. Γιατί εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τη μία ή την πολλαπλή χρήση. Εγώ προσωπικώς δεν έχω ζήτημα για το πώς θα το χειριστούμε το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει σήμανση προϊόντος μίας χρήσεως και γίνεται η επανεπεξεργασία του ε, άπειρες φορές, άπειρες φορές και διατίθεται και πάλι, ο πιο αφελής θα το καταλάβει. Ο κύριος Κάρβανος ε, με πολλή ευγένεια είπε ότι να το πλένουν οι νοσοκόμες και Μα ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δεν έχουμε ιδέα πώς γίνεται η επανεπεξεργασία αυτών των προϊόντων. Όποιος ισχυριστεί ότι ξέρει τι μοίρα, τι επιφυλάσσει η μοίρα σε ένα ενδοσκοπικό ε, εργαλείο με τη μικροσκοπική κάμερα το οποίο έχει μπει στο στομάχι του ενός και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά σε μία μόνη εξέταση αλλά βέβαια δεν χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν έχει κανείς την παραμικρή ιδέα εάν ξαναχρησιμοποιήθηκε και πόσες φορές ξαναχρησιμοποιήθηκε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε σε όποιον πιστεύει ο καθένας να μην πάθουμε τίποτα. Γιατί οποιαδήποτε μόλυνση μπορεί να μεταδοθεί δεν θα μπορεί κανείς να αποδείξει πώς την έπαθε και δεν θα επιβιώσει ενδεχομένω. Δεν θα μπορεί να τον πιάσει καμία θεραπεία. Γιατί κοιτάμε όλες αυτές τις ενδονοσοκομιακές μολύνσεις, γιατί κοιτάμε αυτή την ε, ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά που διαδίδεται και επεκτείνεται διαρκώς. Εγώ είμαι απλοϊκός άνθρωπος κυρίες και κύριοι. Όταν κάτι μου λέει μία χρήση, εγώ θεωρώ ότι θα είναι μία χρήση. Και κάποιο λέει ναι να μην τα αφήσουμε στη, στα χέρια του παραγωγού. Πολύ καλά, αλλά ποιος θα αυτό η Επιτροπή, εμείς, ο παραγωγός είναι αυτός που θα πει και θα αποδείξει γιατί πρέπει να είναι μια χρήση και γιατί δεν μπορεί να γίνει επανεπεξεργασία του προϊόντος. Εγώ δεν είμαι αφελής βεβαίως και γνωρίζω ότι πάντα υπάρχει τρόπος να κόβει κανείς παρά, ε, ε, παράδες, το λέω πολύ χιδέα, με συγχωρείτε, αλλά Υπάρχει δυνατότητα για τον παραγωγό να ισχυριστεί ότι είναι μία χρήση το προϊόν και γι' αυτό ανοίγω αυτή τη δυνατότητα. Για να πούμε ότι όποιος είναι σε θέση να πει ότι μπορεί να γίνει επανεπεξεργασία, κάθε νοσοκομεία, κάθε διαδικασία επανεπεξεργασίας ιατρικού υλικού μπορεί να προβαίνει στην επανεπεξεργασία αυτή Και άρα πάβει να είναι μιας χρήσης και δεν έχει την ετικέτα μιας χρήσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να ε, σημαίνεται τίποτε ω μια χρήσεως, αλλά εν πάση περιπτώσει α είμαστε και λογικοί. Όταν ένα προϊόν σημαίνεται ω μια χρήσεως και χρησιμοποιείται πολλαπλώ, ποια, ποια είναι η αξία αυτής της ε, σήμανση τη ετικέτα μια χρήση ένα καλύτερο σύστημα αναζητώ. Αν έχετε εσείς κάτι άλλο να μου προτείνετε, πολύ ευχαρίστω, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο επουδενεί ποτέ με κανένα ε, τρόπο δεν πρέπει να ε, ξαναχρησιμοποιείται και αυτό το οποίο υπό κάποιε τα λοιπά θα μπορούσε. Αυτά στο συγγνώμη που ε, μακρηγορώ. Ναι, η κυρία Μασέ έχει δίκαιο προς την διαφάνεια, έχει ε, απόλυτο δίκαιο. Η κυρία Λεπάζ αλλά και η κυρία Ριβαζή βεβαίω έθιξαν το θέμα αυτό του σκανδάλου ΠΙΠ. Εντάξει, σκάνδαλα πάντα μπορούν να υπάρξουν, γιατί η εγκληματική ενέργεια, γιατί εγκληματική δραστηριότητα αυτό, η εγκληματική ενέργεια διαχέεται πάντοτε με χιλιάδες ακόμη ελεγκτές ε, από οποιαδήποτε υπηρεσία γιατί δεν ξέρω ποια είναι η υπηρεσία αυτή τροφίμων και κτηνιατρική, η οποία ε, ήταν αρμόδια που για του ελέγχου και με ποιο τρόπο ήταν αρμόδια, αλλά αυτό το κρίνει η Επιτροπή. Εν πάση όμω, η προκαταρκτική, πριν από διάθεση δηλαδή στην αγορά επιτήρηση και οι κανόνε σχετικοί είναι τόσο σαφεί και διαφανείς που, μπορούμε να έχουμε, που θα μπορούμε να έχουμε ε, την έγκαιρη προειδοποίηση ε, και όπως είπα, στο τέλος θα πρέπει να δούμε ποιος θα πληρώνει το λογαριασμό. Δεν θέλω να είναι τα κράτη-μέλη αυτά και τελικά ο φορολογούμενος που θα πληρώσουν τα σφάλματα του παραγωγού εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτά λοιπόν ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. 13 Μαΐου η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα, ψηφίσουμε στην, θα συζητήσουμε στην Επιτροπή στις 29 Μαΐου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 10 Ιουλίου και κατά πάσα πιθανότητα τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια θα συζητήσουμε την έκθεση. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το δεύτερο μέρος αν θέλετε, το σημείο η έκθεση του κυρίου Λίζα, έχετε πέντε λεπτά να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές. Συναντηθήκαμε ήδη πάρα πολλές φορές, ήταν πολύ επικοδομητικές αυτές οι συναντήσεις. Η συνεισηγητρία του, των σοσιαλιστών είναι η κυρία Ροτ Μπέρεντ και αυτό μας διασφάλισε κάποια συμφωνία, κάποια κοινή πλεύση ως προς τις δύο αυτές παρόμοιες εκθέσεις. Λοιπόν, για περί τίνος πρόκειται. Ας το εξηγήσω και εκείνους που δεν ήταν εδώ την προηγούμενη φορά. Τα in vitro διαγνωστικά άλλα, τα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται απευθεία στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αυτών των εργαλείων, για παράδειγμα μέτρηση ε, του επίπεδου γλυκόζης, ε, τεστ για τον ιό HIV... και άλλα τέτοια πολλά προϊόντα. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι τα in vitro διαγνωστικά είναι λιγότερο σημαντικά. Αλλά εγώ έχω να πω ότι πιστεύω πως δεν είναι η μικρή αδελφή, αλλά οι γονείς των ε, ιατροτεχνολογικών προϊόντων εν γέννη τα in vitro διαγνωστικά, διότι χωρίς μια σωστή αγωγή, χωρίς ένα μάλλον ε, σωστό και διαγνωστικό εργαλείο, η αγωγή δεν μπορεί να γίνει σωστά. Πρώτα λοιπόν γίνεται η διάγνωση και μετά δίδεται η αγωγή στην ιατρική. Γι' αυτό λοιπόν η σειρά είναι αντίστροφη πιστεύω. Και εδώ υπάρχουν τα ίδια προβλήματα με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Υπάρχουν ε, τεστ, τέτοια διαγνωστικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, όμως είναι χαμηλής ποιότητας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν τεστ για HIV, για παράδειγμα, που δίνουν ψευδή αρνητικά αποτελέσματα, ενώ ο ασθενής έχει τον ιό HIV. Φανταστείτε λοιπόν τις συνέπειες που έχει μια τέτοια λάθος διάγνωση. Ε, μια εμπειρογνώμονας έκανε μελέτες και μας είπε ότι έκανε ε, ένα τεστ ε, DNA με ένα από αυτά τα προϊόντα, το έστειλε σε τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια και πήρε τέσσερα διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης, σε ανίατες ασθένειε, όπως η πατήτη δασέ, υπάρχουν και εκεί χαμηλής ποιότητας διαγνωστικά προϊόντα. Διεξήχθη συζήτηση και ο συναδέλφος Άμπανοφ είπε ότι πρέπει να προσέξουμε την αρχή της επικουρικότητας εδώ στην έκθεση είναι κοινό λοιπόν έργο, ευρωπαϊκό έργο. Αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Τώρα, όπως είπε και η κυρία ε, Ροτ Μπέρεντ στην προηγούμενη έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σημαντικές ε, βελτιώσεις με την ε, αυτή πρόταση. Πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά βήματα μπροστά, εάν εφαρμοστούν όλα αυτά που έχει προτείνει η Κομισιόν. Υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε κάνει προτάσεις. Σημερίζομαι πολλές από τις προτάσεις της κυρίας Ροτ Μπέρεντ, όπως για παράδειγμα την ποιότητα των κοινοποιημένων οργανισμών. Πιστεύω πως ανεβάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πραγματικά σε αυτό το σημείο συμμερίζομαι και την κριτική που άσκησε η κυρία Ροτπέρεν στην πρόταση. Τώρα όσον αφορά το διάστημα των τριών ετών. Ε, αυτό δεν αφορά την ε, αδειοδότηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Δεν θέλω να σας ε, παρουσιάσω μια τρομακτικά σενάρια. Η παρατήρησή μου όσον αφορά τα τρία χρόνια είναι ότι ε, αρχικά χρειάζεται να εφαρμοστεί νέα νομοθεσία. Η Κομισιόν προτείνει τρία χρόνια για τα ιατροδιαγνωστικά προϊόντα ε, και για τα in vitro πέντε. Εγώ ε, προτείνω να το επιταχύνουμε αυτό έτσι ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες. Εάν όμως τώρα αρχίσουμε από την αρχή τη δημιουργία νέων οργανισμών, τα τρία χρόνια δεν θα μας φτάσουν για να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και σωστά και θα έχει υιοθετήσει και τις βελτιώσεις που έχει προτείνει η Επιτροπή και αυτές που θα προτείνουμε εμείς. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, τις κλινικές αξιολογήσεις, υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως και η κυρία Ροκ Μπέρεντ. Α, επίσης, ε, Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, συμφωνώ επίση και για τις ε, προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή συζητώ με τους ε, συνεισηγητές για τις ε, κλινικές δοκιμές, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις προτάσεις μας από κοινού. Προτείνω μία ρύθμιση για τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, την εξής, την μετάφραση για παράδειγμα της δήλωσης συμμόρφωσης για που θα προορίζεται για τους ε, ασθενείς ή τους χρήστες τέλος πάντων αυτών των προϊόντων να μην μεταφράζεται σε όλα τα κατημέλη, σε όλες τις γλώσσες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν αυτές οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ένα άλλο ε, θέμα πολύ αμφιλεγόμενο είναι, τα, είναι οι εξετάσεις οι ενδονοκλινικές Όσον αφορά αυτό, αυτή τη στιγμή διεξάγω συζητήσεις με πυρογνώμονες και του συνεισηγητές. Έχω μία αρχική πρόταση. Ε, οι επιστήμονες και οι ερευνητέ δηλαδή που ασχολούνται με, κάποια συγκεκριμένη, με κάποιο συγκεκριμένο τομέα να κάνουν εκείνη, λοιπόν που να αρμόδιοι τις κατάλληλες προτάσεις όμως να μην αφήνουν το προϊόντα τελείως εκτός ρύθμισης να κυκλοφορούν στην αγορά. Επίσης, πιστεύω πως χρειάζεται, χρειάζονται πολύ πιο αυστηροί κανόνες για τους συνοδούς διάγνωσης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ε, πολλά ε, διαφορετικά ε, τεστ στο εμπόριο, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ευέλικτη. Μία εταιρεία, για παράδειγμα, που φέρνει στην αγορά ένα προϊόν, πρέπει εκείνη, πιστεύω, να είναι η αρμόδια που θα θέσει τις ε, προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος αυτού. Τώρα, υπάρχει πίεση χρόνου. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, παρουσιάζει μια σειρά πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Και εδώ πιστεύω πως πραγματικά δεν χρειάζεται αυτό, αλλά είναι απόφαση. Ο Επίτροπος Μπόλς, ο οποίος είναι ο αρμόδιος, με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων του, σίγουρα υποστηρίζει την πρόταση των πράξεων κατά την εξουσιοδότηση και δεν θα είναι τόσο ευλίγιστος. Όμως ε, θα έχουμε σύντομα μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως να αλλάξουν τα πράγματα. Ε, και ελπίζω είναι πρόταση να μην έχει τόσο αυστηρές ε, διατάξεις και προδιαγραφέ, ώστε να γίνει η κυκλοφορία των προϊόντων αυτή πιο δύσκολη, αλλά να διατηρήσει τα βασικά στοιχεία και να μην τα αλλάξει μέσω τη επιτροπολογία και των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, αλλά να ακολουθήσουμε την οδό τη συναπόφαση. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ πιο γρήγορο από ότι ε, ένα κανονισμό. Τώρα τέλο. Κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι η συγκατάθεση μέσω, ε, μετά από ενημέρωση. Έχω συζητήσει με εμπειρογνώμονες από τον ΩΣΑ, από το Συμβούλιο, ε, με, με ειδικού ε, γενετιστές και πιστεύω πως ειδικά στην περίπτωση των τεστ DNA είναι πολύ σημαντική η πρώτερη συμβουλή. Διότι αυτά τα τεστ καθ' αυτά είναι σημαντικά. Πιο σημαντικό όμω είναι το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε στο διαδίκτυο, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολλές μη σοβαρέ ε, προσφορέ τέτοιων ε, τεστ και έχουν, μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειε αν αυτά χρησιμοποιηθούν λάθος. Φανταστείτε δηλαδή, σε παρά... για παράδειγμα, έναν εργοδότη, δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο, να συλλέγει γενετικό υλικό, μία τρίχα, να το στέλνει σε ένα εργαστήριο και να αποκτά λοιπόν γενετικές πληροφορίες για τον ενδεχόμενο τον υπάλληλό του, για γενετικές ασθένειες, για κληρονομικές ασθένειες για παράδειγμα. Εδώ πιστεύω ότι χρειάζεται καλή ενημέρωση, σωστή ενημέρωση. Και πρέπει εμείς στο Κοινοβούλιο να την αποφασίσουμε, να την ψηφίσουμε. Τις λεπτομέρειες θα τις επεξεργαστούμε. Ε, πρόταση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται από μένα και από μια ομάδα νομικών και εμπειρογνωμόνων. Ε, προτείνω να ακολουθήσουμε την αρχή που υπάρχει και στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις συνέπειες που έχει η μη σωστή πρώτερη ενημέρωση. Και πιστεύω πως αυτή η βάση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά προς το παρόν. Να σας ευχαριστήσω για την συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Κύριε Ελίζα, είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσουν να συνεννοηθούν οι εισηγητές την επόμενη φορά ως προς τη σειρά των θεμάτων του στην ημερήσια διάταξη για να μην έχουμε διαφωνίες τέτοιου τύπου. Και σας ευχαριστώ μεταξύ και τους δύο. Και τώρα προχωρούμε στους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Ντάτμαντουρ, Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε πολλά από τα όσα μας είπε ο εισηγητής, ο κύριος Λύσε, συμφωνώ μαζί του. Στο θέμα που αφορά την πρόταση Επιτροπής. Νομίζω ότι τα κατάφερε καλύτερα η Επιτροπή αυτή τη φορά. Συμφωνώ σε πολλά σημεία με την πρόταση της Επιτροπής. Και ίσως, κοιτώντας τα ε, τους οργανισμούς αυτούς, το notified bodies, θα πρέπει να δούμε αν χρειάζεται να αλλάξουν οι διαδικασίες ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα και βέβαια η χρηματοδότηση. Στο σημείο που ανέφερε ο κύριος Κλίσε, ναι, συμφωνώ μαζί του ότι η ποιότητα των ε, οργανισμών αυτών ε, πρέπει να ε, βελτιώνεται των κοινοποιημένων φορέων. Ε, πρέπει να υπάρχει η κοινοποίηση, η καλύτερη γνώση του ποιο οργανισμό έχει δώσει ποια άδεια. Δεν μπορεί αυτό να δίδεται δηλαδή σε εργολάβου, σε ιδιωτικέ επιχειρήσει ή ε, κάποιο μεμονωμένο γιατρό ενδεχομένω που κάνει μια ε, κλινική μελέτη. Στο θέμα του χρόνου νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κύριο Όλη, μπορούμε να παρακολουθήσουμε παραλλήλου τα θέματα, να συντονιστούμε για τις καθυστερήσεις που ανέφερε ο κύριος Λίτς. Το επεσήμανα και νωρίτερα, πως είμαι πεπισμένος ότι δεν οδηγεί σε καθυστέρηση ως προς τη θέση στην αγορά ενός προϊόντος η εισαγωγή και μόνο μίας διαφορετικής διαδικασίας από αυτή που ισχύει μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο και να μην έχουμε και καθυστερήσεις. Μπορεί να είναι καλύτερο και να μην έχουμε και καθυστερήσεις στα επιμέρους ζητήματα για τις ε, ενδονοσοκομιακές δοκιμές, ε, και τη διαγνωστική. Δεν είμαι 100% σίγουρη, δεν είμαι πεπισμένη, αν, έχω κατάλαβει καλά, ότι η παρέκκληση την οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένες ενδονοσοκομιακές ε, δοκιμές και κυρίως τη συνοδευτική διαγνωστική, companion diagnostic δεν είναι αρκετά καλές και ότι χρειάζεται προσαρμογή. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον εισηγητή πιο λεπτομερώς, γιατί δεν έχω πιστεί. Ο κύριος Λίζε μας λέει ότι θέλει την προσαρμογή των ενδονοσοκομιακών δοκιμών, αυτών δηλαδή που διεξάγει ένα οργανισμό στο ιστορικό του, ένα φορέα στο ιστορικό του, κάνει τι σχετικέ προτάσει του για τη συνοδευτική ε, διαγνωστική, τα δοκιμές α, για συγκεκριμένους ε, ασθενείς. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά πάντως για τα ε, A-test, για τα κύρια τεστ, για τις κύριες δοκιμές ε, τύπου α, τις συνοδευτικές, νομίζω ότι μπορούμε να συναντηθούμε με τον κύριο Λίζε και να βρούμε καλές λύσεις. στο πεδίο εφαρμογή, που δεν έθιξε ο κύριος Λίζα. Βλέπω πως θεωρεί ότι έχει λησμονήσει, έχει παραμελήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το πεδίο εφαρμογής τις ε, γενετικές δοκιμές. Πρέπει να πω ότι έχω σοβαρές αμφιβολίες ως προς αυτό, αν θα πρέπει δηλαδή να περιληφθεί, για τις ε, πράξεις στην νομοθετική διαδικασία. Είμαι η τελευταία η οποία θα υποστηρίξει την, ε, ή που υποστήριξε ποτέ στο παρελθόν την επιτροπολογία. Ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε με πολύ μεγάλη προσοχή μεριμνούσαμε ώστε να μην μπαίνει ούτε μία γραμμή στην επιτροπολογία η οποία θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγέ στο νομοθέτημα, ε, στην νομοθεσία. Πάντα είναι εκτεριστικέ δηλαδή πρέπει σωστά. Τώρα έχουμε μετά την συνθήκη τη Λισαβόνα, την νομική αυτή βάση που μας επιτρέπει εμένα τουλάχιστον να προχωρήσουμε γρήγορα χάρη στι κατεξουσιοδότηση στην πράξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ δεν έχω καμία δυσφορία στην υπόθεση αυτή. Είναι ακριβώ αυτό το σημείο στο οποίο βλέπω να έχει νόημα η διαδικασία των κατεξουσιοδότησεων πράξεων γιατί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι ένα νομοθέτημα ακόμη και με τρία άρθρα μόνο περίπου 1,5, ένα χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να ολοκληρωθεί μέσα από τη διαδικασία την νομοθετική να περάσει από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο να, ε, ε, να διανεμηθεί στην Επιτροπή να γίνει η ε, διανομή των εκθέσεων και και ούτω καθεξής και μετά οι με τις προθεσμίες για τις τροπολογίες, τη σύνταξη κτλ μπορεί να κρατήσει από 9 μέχρι 12 μήνε η ολοκλήρωση τη διαδικασία αυτή για το Κοινοβούλιο και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πολύ βραδία η διαδικασία και είναι φορέ που χρειάζεται να μπορούμε ταχαίω να αντιδράσουμε, πολύ ταχύτερα δηλαδή σε, με βάση ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ λέω, εκεί που χρειάζεται ευελιξία, εκεί που χρειάζεται ταχύτητα, για το συμφέρον του ασθενού, για συγκεκριμένα ιατρικά προϊόντα, θεωρώ ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη λύση των κατεξουσιοδότησων πράξεων εφόσον τηρείται σωστά η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Τάιλερ. Τέιλορ. Good morning, Καλημέρα σας. Θέλω πρώτα πολύ όλα να ευχαριστήσω τον Δ. Αλίζα για το σχέδιο έκθεσης. Έκανε και σειρά αλλαγών στην πρόταση κομισιών που βελτιώνουν την πρόταση. Υπάρχουν κάποια σημεία για τα οποία δεν είμαι πολύ σίγουρη κατά πόσον κινούσε στην κατεύθυνση. Βλέπαμε το σκεπτικό σα και κάποιε αλλαγέ ακόμη περιμένουμε. Θέλω να αφαιρθώ σε τρία σημεία γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Σε ό,τι αφορά τι κλινικέ αποδείξει, κατανόηση γιατί θέλει να διευκρινίσει τη δομή τη πρόταση Κομισιόν προκειμένου, δίνοντα κάποια κρίσιμα ε, στοιχεία τη πρόταση των κλινικών δοκιμών Κεφάλαιο 6 και παράρτημα 8. Θέλουμε κάποιες περισσότερες εξηγήσει και διευκρινήσεις εν προκειμένου. Θέλουμε έναν τομέα ιατρικών ε, απασχολούμενων στον τομέα της υγείας όπου να μπορούν να λαμβάνουν ημερωμένε αποφάσεις. ό,τι αφορά τις αλλαγές στο τομέα της παρακολούθησης και επαγρύπνησης και την ανάγκη της έγκρισης από κώδικα διοντολογίας είναι κάτι θετικό, περιμένουμε λεπτομέρειες. Έπειτα, χαιρόμαστε γιατί διατηρείται το πυρήνα ε, της προσκοπησιών και μία έγκριση πριν τη θέση στην αγορά δεν θα είναι μια καλή λύση. Τώρα, κάποιε άλλε ανησυχίε ε, για τα περίπτωση τη πρόσβαση, ε, γιατί μάλλον την εξαίρεση in-house. Εκεί μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα για, κάποιες, για κάποια προϊόντα ιδίως όταν είναι, ε, μπορούν να εκτεθούν σε παράγοντες τέτοιους που μπορούν να δημιουργήσουν θανατηφόρες λοιμώξεις. Μόνο όταν τα πρώτα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν ε, εμπορικά και για πολύ σπάνιες ε, νόσους και για ένα ποσοστό ασθενών πολύ πολύ χαμηλό θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιων νόσο που απαιτούν άμεση ε, επίσης ε, νοσηλεία και θεραπεία. Είναι περιπτώσεις που μπορούμε να δεχτούμε ε, πιο χαλαρούς κανόνες. Το τρίτο ζήτημα που θέλω να αφαιρθώ είναι ο αυτοέλεγχος. Εκεί τίθεται ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη διάγνωση νόσων που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη ψυχολογική πίεση του ασθενούς. Δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι, έχει νόημα να βάλουμε τέτοιου κανόνε σχετικά με τον αυτοέλεγχο και το γενετικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι η σε αρχή επικουρικότητα είναι καλό τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν κατά πόσον μπορούν να απαγορεύουν κάποιε τέτοιε δοκιμέ. Και επειδή απαιτεί και η διαδικασία τη συνένεση για του αυταελέγχου, τίθεται θέμα εθνική κυριαρχία, για παράδειγμα. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητείται και η συνένεση και για παιδιά κάτω από κάποια ηλικία. Στο συγγνώμη αν ε, τρέχω, αλλά προσπαθώ να κρατήσω το χρόνο, κάτι άλλο. Πώς ορίζεται ε, αυτό το προϊόν στο κείμενο. Είπατε ότι μιλάμε για δοκιμέ για τον κύκλο ζωή ε, και είναι προϊόντα που έχουν άμεσα ή έμεσα η εμεσα η στο τομέα της υγείας. Προσπαθώ να δώσω τον ορισμό με μεγάλη προσοχή και πιστεύω το σκεπτικό να καλύψουμε και τι δοκιμέ που μπορούν να καθορίσουν την προδιάθεση των ασθενού, ε, την γενετική προδιάθεση για μία ασθένεια, είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Πρέπει να διευκρινίσουμε ποιε είναι οι συσκευέ εκείνε που μπορεί να καθορίσουν προδιάθεση ή κίνδυνο για μη ε, θανατηφόρα ε, ασθένεια ε, γιατί αυτό σχετίζεται και με το πώς θα ορίσουμε στο μέλλον πιθανές ε, ασθένειες που, για τις οποίες κινδυνεύει και η ίδια η, ζωή. Κύριε Άλπεν, ευχαριστώ Ματίας που μου δίνετε το λόγο. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτερ Λίσσα για την εξαίρετη δουλειά του και για την δυνατότητα που μας, έφερε, που μας έδωσε να συμμετέχουμε πλήρως στην προετοιμασία της εκθέσεως. Υπήρξαν κάποια σημεία αρκετά απλά, αλλά κάποια άλλα ήταν πάρα πολύ περίπλοκα και γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερως μας επέτρεψε να συμμετάσχουμε πλήρως στην προετοιμασία. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία λοιπόν που πρέπει να προβάλλουμε ιδιαίτερως εμείς. Το self-testing. Αυτό εξέτασε και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις. Πρέπει να διαφοροποιηθούν. Χρειάζεται μια πολύ πιο συγκεκριμένη διάκριση. Ο ασθενής πρέπει να συνοδεύεται από πιο πολλές ε, πληροφορίες, συμβουλές ούτω υπήν όταν ξεκινάει την αυτοεξέταση. Δεν νομίζω να διαφωνεί σε αυτό ο κύριος Λίζα, άρα χρειάζεται να ενισχυθεί η υποχρέωση εξήγηση. Ο κύριος Λίζα, επίσης, βλέπω θέλει να αναβάλει την ε, υλοποίηση. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. Είχε αρκετό περιθώριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία. Η κυρία Ροτμπέρεντ το επεσήμανε ήδη. Έχει δουλέψει καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει δείξει την απαραίτητη επιμέλεια. Η ενεπιγνώση συνένεση τώρα ε, συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση και θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτή τη δέσμευση που περιλαμβάνεται στο χάρτη των δικαιωμάτων των ασθενούς, του ασθενούς όπως άλλωστε και για τις ε, κλινικές δοκιμές ε, αναφέρεται ότι απαιτείται η ενεπιγνώση συνένεση και εμεί αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Πολλοί σας μιλάνε για διαφάνεια. Γίνεται πια αυτή η διαφάνεια ε, μια εποδός που ίσως κουραζόμαστε να ακούμε. Αλλά η διαφάνεια που χρησιμοποιείται διαπάνω των επιστητών έχει στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση κέρια σημασία. Έτσι ώστε τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην αγορά, να φτάνουν στην αγορά χωρίς τα κρυφά ελαττώματα ή χωρίς την ενδεχόμενη, όπως λέμε, απόκρυψη κάποιων στοιχείων, εκεί που δεν μας λένε τα πάντα. Πρέπει δηλαδή να είναι ο ενδιαφερόμενος εν γνώση, ο ειδικό ιδιαίτερο να είναι εν γνώση όλων των στοιχείων, ώστε να μπορεί να προλαμβάνει και όχι να θεραπεύει. Ξέρουμε ότι πάντα προκαταρκτική διάγνωση ίσως είναι πιο δύσκολη, αλλά όπως είπε η κυρία Ροτσβέρεντ, αν, αν αποφύγουμε τα κενά, τα ε, χάσματα στην νομοθεσία, τα loopholes όπως τα είπε, νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά αυτό το θέμα της ε, διαγνωστικής in vitro. Είναι πολλοί γιατροί που δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες. Και εμείς ακόμη στη Δανία που έχουμε πολύ μεγάλη ε, διαφάνεια, όπως και στη Γερμανία που ξέρω ότι είναι και επιφυλακτική οι γιατροί πολλοί είναι επιφυλακτικοί γιατί διότι φοβούνται αυτές τις δοκιμές, αυτά τα τεστ ε, ή τις θεραπείες ακόμη για τα οποία δεν έχουν πλήρη στοιχεία. Άρα χρειαζόμαστε πιο πολλά στοιχεία, πιο γρήγορες διαδικασίες, αλλά και πιο διαφανείς και βέβαια θέλουμε την δότηση πριν από τη διάθεση στην αγορά για τα προϊόντα ε, που μπορεί να ε, επιφέρουν κινδύνους. Αυτό πρέπει να οριστεί υποχρεωτικά, να μην μπορεί κανείς δηλαδή να αποφύγει την αποκάλυψη στοιχείων αποτελεσμάτων δοκιμών ενδεχομένω που εστέθησαν με αποτυχία. Δεν μπορεί δηλαδή να προβάλλονται μόνο τα θετικά αποτελέσματα. Για τους ε, κοινοποιημένους φορείς. Αρκούν αυτοί, αποτελούν επαρκή εγγύηση όταν έχουμε ένα κεντρικό σύστημα, ένα κεντρικό όργανο για τους ελέγχους. Να σας πω, υπάρχει εδώ ένα παράδοξο, ένα οξύμορο ή καλύτερα ένα δίλημα μεταξύ της ταχύτητας και της διαφάνειας. Ε, Βεβαίω, εγώ προτιμώ πάντα τη διαφάνεια. Αλλά όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και όταν έχουμε κοινοποιημένου φορεί οι οποίοι δεν είναι καλά ενημερωμένοι και πληροφορημένοι. Σε τι βελτιώνεται η ασφάλεια. Ε, τότε ας έχουμε καλύτερη διαφάνεια για να μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις οι οργανισμοί αυτοί. Κύριος Κάρμπανοχ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομο. Να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή, να τον ευχαριστήσω και για την συνεργασία με τους κοιόδη εισηγητέ. Οι προτάσεις του βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητή είναι υπέρ μια αργής μετάβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Όπως και στην προηγούμενη έκθεση, πρέπει να βρούμε μια εξισορροπημένη θέση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ποιότητα από τη μία και την προσβασιμότητα στην ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την άλλη. Εάν εμείς, υποστηρι... Ε, εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε μια... Ε, έναν εξυγχρονισμό της... των ιατρικών υπηρεσιών. Τότε, λοιπόν, πρέπει να υποστηρίξουμε τις κορυφαίες ιατρικές ε, υπηρεσίες και στα κέντρα εφαρμογής τους και επίσης την προληπτική φροντίδα σε πρωτογενές στάδιο πρόληψης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω για παράδειγμα να κάνουμε διαγνωστικά τεστ, να κάνουμε screening ε, στους ε, ασθενείς. Και επίσης μια άλλη σειρά δοκιμών κατευθείαν στα ε, ιατρία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την συζήτηση για αυτό το θέμα και έχει το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για την εντότητα που μας δίνετε να ακούσουμε τις απόψεις Συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπατε. Ανεξάρτητα με τη σειρά με την οποία τα σημεία, είναι εξίσου σημαντικά, εξίσου σημαντικές προτάσεις και έτσι και εμείς τα είδαμε και τα προσεγγίσαμε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα πολλά από τα σημεία ε, που επεσήμανε και ο εισηγητής και οι σκιώδες, εγώ θα εστιάσω σε αυτά που φαίνεται να ε, γίνουν περισσότερη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα για τους ε, φορείς κοινοποίησης, ο κύριος Λύς ε, το ίδιο πράγμα το είπαμε και πριν για την προηγούμενη πρόταση. Για να είμαστε σίγουροι ποιε είναι οι τάξει που να εφαρμόσουν σε αυτό το τομέα και εμεί το προσέχουμε για τι κλινικέ δοκιμέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είπατε ότι συνεργάζεστε και με τον εισηγητή και την πρόταση, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση. Ό,τι προβλέπετε σε μια πρόταση να μην έρχεται σε σύγκρουση με την άλλη. Για το πολύ ευαίσθητο ζήτημα που θέσατε τώρα. Για τη συνένεση μετά από ενημέρωση ιδίως ε, για τεστ όπως ε, αυτό του DNA που είναι πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι και εμείς σε αυτό το τομέα και οποιαδήποτε βελτίωση μπορεί να γίνει σε αυτό το τομέα πραγματικά είναι κάτι που χαιρετίζουμε. Θέλουμε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Καθώς βλέπουμε ότι στο μέλλον μάλλον θα είναι όλο και πιο συχνά αυτά τα τεστ. Σε ό,τι αφορά τα τεστ που γίνεται in-house, κατανοώ αυτό προτείνει ο εισηγητής να υπάρχουν οι κατάλληλες απαιτήσεις που θα εφαρμόζονται πάντως ότι αφορά για αυτά τα τεστ κύκλου ζωής, ναι, από τη μία πλευρά κατανοούμε την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις, δηλαδή ε, ποια τεστ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και υπό, και υπό τον ορισμό του ε, ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Μεταβατικές περίοδοι. Θέλουμε συντομότερες μεταβατικές περίοδους ώστε η νομοθεσία να εφαρμόσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει ορθά. Η διατήρηση της περίοδου 18 μηνών ε, για την καταχώρηση των ε, οικονομικών φορέων, προϊόντων και πιστοποιητικών είναι κάτι πολύ σημαντικό αν βραχυνθεί μεταβατική περίοδος, τελικά, να είμαστε σίγουροι ότι δεν κινούμεθα κατά του ίδιου μας του σκοπού. Θα πρέπει να έχουμε και έτοιμα τα πρακτικά μοντέλα όταν θα αρχίσει να εφαρμόσετε η πρόταση. Στο λέω, με το λάβετε και αυτό υπόψη, για τις πράξεις και την εξοδότηση. Ένα σχόλιο. Πάντοτε θέλουμε να διασφαλίσουμε την ακολουθία στην Κομισιόν δεν αποκλείουμε ποτέ από αυτό που ε, καταρχήν ε, συμφώνησε ο νομοθέτης ή οι νομοθέτες. Σίγουρα θέλουμε να διασφαλίσουμε την ακολουθία. Κάποιες φορές η πρακτικοσοδότηση ακολουθια καποιες φορες η εισοδοτηση κινουνται πιο γρήγορα από ό,τι στην απόφαση. Θα στο λέω, αλλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσετε εσείς οι νομοθέτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιταλίζα να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, συνησυγητέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σύντομα να πω ότι πολύ σωστό αυτό που είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ για τα ενδοκλινικ... τις ενδοκλινικές δοκιμές. Πρέπει να το δούμε. Έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ελαττωθεί η ασφάλεια, αλλά όμως εάν η βιομηχανία δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει να κυκλοφορεί στην αγορά ασφαλή προϊόντα, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα ε, νοσοκομεία, έτσι ώστε να δοθούν οι δυνατότητες αυτές. Έχουμε πολλές ε, απόψεις για το θέμα αυτό και πρέπει να τις ε, συνενώσουμε, όπως είπε και η Ρεμπέκα. Σύμφωνα με αυτό, άλλες απόψεις επίσης ε, ίσως πάνε λίγο πολύ μακριά και πρέπει να τις επεξεργαστούμε. Όσον αφορά το, το πεδίο εφαρμογής δεν έχω να πω κάτι. Πιστεύω πως η Dagmar Rothberg και οι άλλοι έχουν αναφερθεί εκτενέστατα σε αυτό, είναι δύσκολο να πούμε τι γίνεται σε περίπτωση ενός τεστ το, οποίο θα το πώς θα εφαρμοστεί μάλλον ένα τέτοιο τεστ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιο θέλει να χάσει βάρο και χρησιμοποιήσει ένα τεστ που θα τον κάνει να αποφασίσει αν θα κάνει δίαιτα και ποια θα είναι αυτή ή όχι. Αυτό είναι κάτι που ε, εξαρτάται από τον ασθενή. Αν ο ασθενή πρέπει οπωσδήποτε συντομότατα να χάσει βάρο, τότε σίγουρα εάν το τεστ δεν είναι καλό, δεν είναι κατάλληλο και η δίαιτα αυτή που θα ακολουθήσει ο ασθενή δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική βάση, αλλά είναι τελείω αυθαίρετη, τότε φυσικά αυτό είναι εξίσου προβληματικό ε, με άλλα τεστ τα οποία δεν ε, υπόκειται σε κάποια ρύθμιση. Τώρα, το πού αρχίζει η ιατρική, πού τελειώνει η ιατρική με αυτά τα προϊόντα είναι κάπως ασαφές. Πρέπει να προσέξουμε και να προσαρμοστούμε στον κανονισμό και να τον προσαρμόσουμε ανάλογα. Τώρα, όσον αφορά την ενημερωμένη συγκατάθεση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη ορισμένους εισηγητές και την Επιτροπή. Η Ρεμπέκα Τέιλο ρώτησε εάν αυτό υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ή στην αρχή της επικουρικότητας. Ναι, το κατανοώ αυτό. Ο, κρατανοώ το ότι προέρχεται από το Ενώμενο Βασίλειο ε, αυτό, αυτή η ερώτηση. Εάν με ενημερώνει καλά η νομική μου υπηρεσία, αυτό δεν αναφέρεται στο άρθρο 3. Είναι μια αρχή την οποία έχουμε αποφασίσει από κοινού, είναι νομικά δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζεται στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνει υπόψη αυτές, και εμείς λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις αρχές. Όταν υπάρχει νομική βάση, τότε υπάρχει και η δυνατότητα, όχι μόνο η δυνατότητα μάλλον, αλλά και η υποχρέωση να υπάρχει ενημερωμένη συγκατάθεση, το informed consent. Και αυτό πρέπει να το πράξουμε κιόλα. Φυσικά, εντάξει, μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και να καμφθούμε κάπως σχετικά με τη διατύπωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γενετικά τεστ, τα οποία διεξάγονται στα πλαίσια μιας φυσιολογικής αγωγής ή μιας διαγνωστικής θεραπείας ή έχουν ζητηθεί από έναν γιατρό για να αποφασίσει τι αγωγή θα ακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα τεστ έχουν συνέπειε. Δηλαδή, δεν άμα κάνει ας πούμε, ένα ένα τέτοιο τεστ και του πούνε ότι στα 50 σου θα πάθει αυτή την ανίατη κληρονομική ασθένεια, είναι τρομακτικέ οι συνέπειε. Πρέπει να τι αναλογιστούμε. Τώρα, όσον αφορά τη διαφάνεια, ναι, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ανάλογους, ε, ανάλογες ρυθμίσεις ε, με τις κλινικές δοκιμές. Και ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο που μου επέστησε την προσοχή τη, στην σημασία και στο ειδικό βάρος που θα δώσουν οι εμπειρογνώμονες σε αυτή την έκθεση. Τώρα το πώς θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια ή τουλάχιστον την ε, ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Ε, στο εργαστήριο του ε, Dennis Filmes, όπου ήταν παρόντες και επιρρογνώμονες από το Ιατρικό Ινστιτούτο, είδαμε ότι μπορούμε, για παράδειγμα, σε ασθενείς με μία σπάνια ασθένεια, χρησιμοποιώντας αυτές τις δοκιμές, προστατεύοντας και τα προσωπικά τους δεδομένα, να μάθουμε πάρα πολλά. Τώρα η Μάγκαρα Τάουκιν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και το 2011 είχαμε ήδη συζητήσει. και Ήταν κυρία Ροτ Μπέρεντ εκεί για το, πώς, για το ποια τακτική θα ακολουθήσουμε και πραγματικά ούτε εγώ θέλω τα δεδομένα των ε, ασθενών να χρησιμοποιηθούν, να κλαπούν για περιεργού σκοπούς. Πραγματικά πιστεύω πως η δουλειά που κάνουμε στην προστασία δεδομένων και στην προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων είναι πολύ καλή Χρειάζεται, ναι, βέβαια, να ενισχυθεί. Πρέπει να τηρείται η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων και να αποφεύγεται να αποφεύγονται οι αρνητικέ συνέπειε και οι ζημιέ του ασθενεί εάν τα δεδομένα αυτά δημοσιευθούν και πιστεύω πω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά αυτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λίζα. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, και στις 29, όπως και για την έκθεση Ροτ Μπέρεντ, συζήτηση με τις τροπολογίες στην Επιτροπή, ψηφοφορία στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ολομέλεια ενδεικτικά προβλέπεται τον Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ όλους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα έκθεση Κράμερ. Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Όσοι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη συζήτηση παρακαλώ να αποχωρήσουν. Βεβαίω, όποιο θέλει να παραμείνει είναι ευπρόσδεκτο, αλλά παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχω. Ο εισηγητή τώρα μπορεί πολύ γρήγορα να αναλάβει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τον λόγο πρόεδρε. Ύστερα από τα όσα ακούσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση δεν είναι δύσκολο να κάνω και εγώ την παρουσίασή μου. Είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα. Έχουμε λοιπόν τη συζήτηση για το recast, για την επαναδιατύπωση. Είχαμε συζητήσει για το πρόγραμμα δράσεως και τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα οχήματα προσωπικής χρήσεως Σήμερα μπορούμε νομίζω να προβλέψουμε που θα εκλειφθεί απόφαση για συμφωνία στο πακέτο για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα με κινητήρα. Κάποια θέματα πιστεύω μπορούν να συμπεριληφθούν στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Δεν χρειάζεται να ξαναρχίσει όλη η συζήτηση του 2009. Μια σύντομη επισκόπηση για τις τροπολογίες. Είναι πολύ λιγότερες από ό,τι περίμενα ή από ό,τι ανέμενα, 120. Μάλλον λίγες μπορούν να κρυθούν για ένα θέμα συγκρινόμενο με τόσο διαφιλονικούμενα ζητήματα. Τα τέσσερα λοιπόν κύρια σημεία των ε, τροπολογιών επικεντρώνονται σε στα έξι στι διαφορέ ανάμεσα στα προσωπικά στα και οχήματα, ε, ε, ε, επαγγελματικά οχήματα και τους ε, στόχους μέχρι το 2020. Επίσης υπάρχει αυτή η, λέξη, αυτή η φράση κλειδί, to be confirmed, προς επιβεβαίωση. Επίσης, μια συζήτηση για το ερώτημα του αν τώρα θα πρέπει να ε, λάβουμε αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά το 2020. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες ε, που υποστηρίζουν άλλες αυστηρές προδιαγραφές από το 2020 και μετά, άλλες από το 2017 και μετά. Επίσης, Πολλές τροπολογίες ε, ε, μάλιστα κάνουν λόγο σε πλήρη διαγραφή του αρχικού κειμένου της Επιτροπής. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πιστεύω πως καλύτερα για οικονομία χρόνου να μην την κάνουμε. Ε, επί, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια, κάποια συμβιβαστική λύση για τον κύκλο δοκιμών των ε, οχημάτων αυτών. Πιστεύω πως θα μπορούσε να προσαρμοστεί με το VENT. Διαφορετικά θα προκύψουν προβλήματα. Βέβαια έχουμε μία πρώτη βάση έτσι ώστε να, να συμβιβαστούμε. Πιστεύω πως μετά από τη συζήτηση θα μπορέσουμε να, να ε, οδηγηθούμε σε συμβασμό πολύ πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Τώρα θα λάβουν το λόγο εκ μέρους του, ΕΦΑ... του ΕΛΚΑ ο κύριος Σοποτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ε, συνεδριάσεων των ε, σκιωδών για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με την έκθεση Όλμερ. Απλά θα ήθελα να πω ο στόχος του 146 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι αδιαπραγμάτευτος όρος. Και πρέπει να πείσουμε όλους τους συναδέλφους προς αυτή την κατεύθυνση. Για τα υπόλοιπα ζητήματα θα είμαι συνεκτικός. Για τα super credits το βλέπετε και σε κάποιες τροπολογίες που ήδη υποβάλαμε. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να δοθούν κίνητρα στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο να σταματήσουν ε, να χρησιμοποιούν τα super credits το 2015. Θέλω να επισημάνω ότι τα εμπορικά οχήματα Ε, η βιομηχανή που με αυτό το κλάδο επενδύει ετησίως 26 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το νέο κύκλο αποδείξεων Κατανοώ τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για να δεχτώ αυτή τη θέση ισχύ ενός νέου κύκλου δοκιμών μάλλον, ως νοοκύκλου δοκιμών για ένα προϊόν που δεν έχει μπει ακόμα στην αγορά και δεν έχουν γίνει ακόμα ε, και τα πρώτα τεστ. Γι' αυτό βλέπετε και σε τροπολογίες που λέμε ότι πρώτα απ' όλα να ο πρώτο κύκλο ε, δοκιμών για το 2017 και άρα ορισμός των στόχων ε, να γίνει για μετά το 2020 βάσει των αποτελεσματών που θα μας δώσει ο πρώτος κύκλος δοκιμών. Κατανοώ τις θέσεις ε, επίσης των σοσιαλιστών και των πρασίνων. Όμως είναι πρόωρο κατ' σήμερα, στην παρούσα κατάσταση, με την κρίση που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητομηχανία, να ορίσουμε τέτοιους στόχους που θα επιτευχθούν το 2020. Αναγκαίο είναι να είμαστε πιο σύνετοι προκειμένου. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε απόψε. Μετά από τις δύο σημαντικές προθεσμίες που σας παρουσίασα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Μαρίτα Όλσκογκ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χόλγκερ Κράμερ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Έχει κάνει μία ακόμα έκθεση σχετική με οχήματα. Δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη έκτακτη συνεδρίαση για να στήσουμε τις λεπτομέρειες, θα το κάνουμε αυτό αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν μου είναι κάπως δύσκολο να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πράγματα που αναφέρονται στην έκθεση για το πού θέλουμε να πάμε. Τώρα, όπως είπε ο κύριος Κράμερ, πρέπει φυσικά να δούμε το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων ε, ξεχωριστά από ότι, ε, τα επιβατικά οχήματα. Δεν είναι τα ίδια. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε μερικά ωφέλη, να βασιστούμε πάνω σε αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί για τα γιοταχή. Για παράδειγμα, αν χρειαζόμαστε έναν κύκλο δοκιμών, ο οποίος θα είναι παρόμοιος τουλάχιστον στο πνεύμα με αυτόν που θέλουμε εμείς για τα επαγγελματικά οχήματα. Επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε την οικονομική κρίση υπεύθυνη για όλα εδώ στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής ε, της κοινοβουλευτικής θητείας έχουμε να, έχουμε να εργαστούμε κάτω από συνθήκες ύφεση, η οποία δεν θα τελειώσει σύντομα, θα διαρκέσει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι εμείς πρέπει να αναβάλουμε τα πάντα ότι πρέπει να σταματήσουμε όλα τα πολιτικά project, ότι πρέπει να ξεχάσουμε οποιαδήποτε πολιτική θέληση. Όχι, πρέπει να ασχοληθούμε μακροπρόθεσμα με το θέμα του περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε καμία παύση, κανένα διάλειμμα των δραστηριοτήτων μας, ειδικά σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι πάρα... Πως, ε, μάλλον με χαρά μου διάβασα όλες αυτές τις ε, τροπολογίες που υποβάλλατε. Είναι αρκετά φιλόδοξες ως προς το περιβάλλον. Τώρα, Πιστεύω πω αυτέ ε, οι προσανατολίε προσανατολίζονται στο τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώ όμω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ χαμηλέ φιλοδοξίε όσον αφορά τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με αυτό που έχει κάνει για τα επιβατικά οχήματα και, το, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώ η πρόταση για αλλαγή για το 2020 και για το 2025 είναι ωστόσο κάτι καλό, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βλέπουμε τι γίνεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τον τομέα των μεταφορών. Αυτές αυξάνονται συνεχώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε την κατάσταση μακροπρόθεσμα. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένους και πολύ στοχευμένους, ε, στοχευμένους στόχους και πρακτικές. Επιπλέον, πρέπει να προσέξουμε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων να αποφύγουμε μία διατύπωση η οποία θα υπονομεύσει οποιαδήποτε φιλόδοξη ε, πράξη της Εκομισιόν. κύριος Κάρλ Σλίτερ. Δεν κατανοώ αυτή την αιμόνη με τα 147 γραμμάρια. Βασίζεται σε λάθος ε, ε, υποθέσεις και σε τελείως διαφορετικό είδος οχημάτων. Το μόνο λογικό θα ήταν η εξοικονόμηση για των ε, χρημάτων και για τον καταναλωτή ε, και για τον κλάδο. Η όλη μελέτη αντικτύπου τι μας δείχνει, ότι θα πρέπει η πρόταση θα πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά με την εξοικονόμηση χρημάτων για την όλη βιομηχανία και τους χρονιτές. Θα θυμάστε αυτή την ε, αυτό που λέμε συχνά ότι στη μία περίπτωση θέλουμε να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο και την άλλη την ευκαιρία. Αλλά ναι μεν υπάρχει κίνδυνο, λένε κάποιοι αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ευκαιρία και μην χάσετε την ευκαιρία μέσα σε μια κρίση. Ε, αυτό είναι μια άποψη, μια θέση που κάποιοι έχουν πολύ ίδιο σε κρίσεις. Μα στην κρίση είναι καλύτερο να επενδύει κανείς γιατί τότε σιγά σιγά θα έρθει η οικονομία και πριν δηλαδή αυξήσουν τιμέ. Στην κρίση λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει τελείω διαφορετική κατάσταση από αυτή που προτείνεται εδώ. Εξοικονόμηση τη εργασία και αύξηση θέσεων εργασία. Ποιο θα αγοράσει εμπορικά οχήματα στο μέλλον αν χρησιμοποιούν ε, δίζελ. Ποιο θα αγοράσει αυτά τα οχήματα το 2025. Αυτά τα αυτοκίνητα ε, στην Ασία θα είναι η καλύτερη αγορά. Εκεί θα σπαταλούν τα χρήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Αν νομίζετε ότι προστατεύεται η βιομηχανία ρίχνοντας τόσο πολύ τα πρότυπα, ε, τότε δεν εξυπηρετείται κανέναν. Σου με τα super credits. Έτσι όπως έχει σήμερα η νομοθεσία, ποιος τα χρειάζεται. κανένα δεν τα χρησιμοποιεί. Γιατί λοιπόν ένα τόσο περίπλοκο χρονισμό με λεκτικά συστήματα, γιατί σπαταλάμε χρόνο και κόπο σε αυτό θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε πιο πολύ τον πύχη της φιλοδοξίας, τότε ναι, θα χρειαζόμασταν super credits. Αλλά έτσι όπως είμαστε σήμερα, και αυτό προτείνουμε, δεν χρειάζονται. Από εκεί πέρα ένα σκάνδαλο. Σε ό,τι λέμε για την κατανάλωση καύσιμο. Παραπλανάται πραγματικά ο καταναλωτής. Αν ο στόχο ειναι είναι μείωση κατά 20-30% των ρήπων, αυτό αντίκειται πλήρω στη λογική τη ενιαία αγοράς. Είναι, υπάρχει απόλυτη παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Εν προκειμένου, ευθύνη δική μας είναι να το διορθώσουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν. Και όπω είπα και πριν, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν κρυφό εργαλείο για να αυξήσουμε αυτόν τον τρόπο τα πρότυπα. Θα πρέπει να αλλάξει ο κύκλος με ορθό τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε να αλλάξει ο κύκλος για να μπορούν οι καταναλωτές να εκτιμούν καλύτερα ε, πόσο τους κοστίζει το καύσιμο καθόλου το κύκλο ζωής του οχήματος. Δεν βλέπω λοιπόν σύγκρουση ανάμεσα στα ε, επιχειρηματικά ε, συμφέροντα, το τι συμφέρει το περιβάλλον και το καταναλωτή. Πιστεύω ότι πάνε παράλληλα αυτά τα συμφέροντα. Γιατί να τα σπαταλάμε αυτά τα χρήματα. Δεν βλέπω όσου είναι και παράξενοι εδώ στο Κοινοβούλιο να θέλουν να αυξηθεί το κόστο για τι επιχειρήσει. Πώ δηλαδή μπορεί αυτό να ωφελήσει τη βιομηχανία. Είναι πολύ κακή η βιομηχανική πολιτική. Παρακαλώ να την καταργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σλίτσερ. Ο κύριος Κάραρον. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με χαρά πάντα ακούω τον φίλο Κάρλ. Αυτή τη φορά δεν θα πω πάλι ως συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελείως λάθος θέση του. Τα επαγγελματικά δεν είναι επιβατικά αυτοκίνητα. Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι για φορτίο, για ε, έχουν ανταλλακτικά, έχουν κομμάτια τα οποία μπορούν να βγουν ή να μπουν. Ε, πολλές φορές τα αγοράζουν μάντρες ε, για να το διαλύσουν και κοιτούν μόνο τι είδους ανταλλακτικά μπορούν να αξιοποιήσουν ή πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν με όσο το δυνατόν ε, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο κόστος τα οχήματα αυτά. Άρα ο παραγωγός ίσως τίνει να παράγει το πιο μικρό ε, επαγγελματικό αυτοκίνητο. Δεν έχει νόημα όμως να έχουμε πάρα πολύ μικρά αυτοκίνητα επαγγελματικά, διότι τότε θα χρειαστεί ο επαγγελματίας να έχει δύο τέτοια ενδεχομένω, χρησιμοποιώντα βέβαια περισσότερα καύσιμα και άλλου φόρου, και ω εκ τούτου δεν είναι πολύ λογικό. Ο κύριο Σλίτερ νομίζω ότι δεν έχει κάνει πολύ λογικές προτάσεις ω προς την οικονομική διάσταση και την περιβαλλοντική τη υπόθεση αυτή. Καταλαβαίνω ότι τον παρασύρουν οι θέσεις και η ιδεολογία του, αλλά δεν είναι σωστέ οι επιλογέ του. Και ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ, τον το Χόλγκερ για την πρότασή του. Ε, είναι σωστή η απόφαση για τα 175 γραμμάρια και τα 147 ως το όριο για το 2020 και συμφωνώ και με την πρόταση του κύριου Ταρταρέλου. Με την έκθεση που είχε από την οποία είχε προκύψει το παράδοξο των 147 στην αρχή. Αυτή είναι η κατάσταση όμως και με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο και έτσι με πολύ οδυνηρό τρόπο φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη που δεν χρειάζεται νομίζω πλέον να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε. Άλλωστε θα υπενθυμίσω ότι ο τίτλος της ε, έκθεσης είναι ο καθορισμός των λεπτομεριών της επίτευξης του στόχου μείωσης. στόχος. Όπως λέει το Υπουργείο Μεταφορών του Ορμένου Βασιλείου, σημαίνει εξοικονόμηση 50 εκατομμυρίων λιρών σε ε, εκπομπές μέχρι το 2032. Άρα οι δύο αυτοί στόχοι που προκύπτουν οι πράσινοι και οι εγκούε, θα έχουν πολύ δυσμενεί συνέπειες και για την βιομηχανία, για τους παραγωγούς, αλλά και για όσους ε, χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά. Και μπορεί ο κύριο Σλίτερ να μην χάρη που θα τα ακούσει, αλλά σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας αναμένεται το 2032 να έχουμε τις χαμηλότερες πωλήσει αυτοκινήτων. Ε, ούτως ή άλλως έχουμε μια σειρά και συνεχίζεται το τσουνάμι του κλεισίματος των εργοστασίων ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Χάνουν οι παραγωγοί χρήματα και ιδιαίτερα από τα μικρότερα οχήματα στην Ευρώπη. Δεν θέλω θα πρέπει λοιπόν να επιδεινώσουμε την κατάσταση αυτή. Για ε, κάποιε από τι επιμέρου πτυχέ τη εκθέσεω. Βλέπαμε χαρά ότι οι παρεκκλήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφυλάσσουν τον απαραίτητο μικρό όγκο, από τον παραγωγό μικρό όγκο από, την ε, ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση. Έχω κάνει τις δικές μου τροπολογίες ώστε να διευρυνθεί η ακουστευμένη προσέγγιση για τους πολύ μικρούς παραγωγούς, παράγουν λιγότερα από 700 οχήματα και που ούτως ή θα έχουν ε, επίπτωση ε, στις συνολικές μειώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, διότι ε, έχουν το 0,21% των ευρωπαϊκών πωλήσεων αυτή η μικρή παραγωγή. Αλλά θα ήταν από την άλλη σωτήριο για αυτούς που προσφέρουν ε, τόσο χρήσιμα έργο παραγωγούς να τους απαλλάξουμε τα 25.000 ευρώ της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Επίσης, Έχουμε καταθέσει τροπολογίες για διαγραφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ε, τη επιβάρυνση για του παραγωγού μα το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο κανονισμό πρέπει να είναι πολύ πιο προσαρμοσμένο στην αναγνώριση και ε, την παρακολούθηση των υφισταμένων συνθήκων όσον αφορά τι δοκιμέ και τις τροπολογίες εκείνε οι οποίε προσπαθούν να εισαγάγουν ε, ένα νέο κύκλο δοκιμών για τα ελαφρά ε, επαγγελματικά οχήματα δυνατό Εμείς αντιδρούμε. Είναι πολύ δεσμευτική αυτή η ώρα των δοκινομών για ορισμένου παραγωγού και μπορεί κάποιοι να προτιμούν διαφορετικούς κύκλους δοκιμών και να αλλάζουν ε, συνέχεια τα δοκάρια του τέρματος ε, προκειμένου να διευκολύνουν τους, ε, τις δικές τους, να προαγάγουν τις δικές τους προτιμήσεις, ωστόσο θα αντιδράσουμε. Εάν η οικονομία παραμένει λοιπόν στάσιμη και αν ε, όπως προβλέπετε βρεθούμε ενώπιον τόσων μεγάλων προκλήσεων δεν πρέπει να εισάγουμε ακόμη πιο αυστηρούς κανόνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Γκόλγκερ για τις ε, προτάσεις του και πάντα είμαι έτοιμος για συνεργασία ώστε να βρούμε μια καλή και ισορροπημένη λύση. Ευχαριστώ. Κύριος Γκρότα. Πριν λάβω το λόγο κύριο ο κύριος Λίτερ θα πάρει το λόγο για ακόμη 25 δευτερόλεπτα. Μια και το όνομά του ακούστηκε τόσες φορές θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Και βλέπω ότι ο κύριος Κάλαναν γελάει ικανοποιημένο. Αγαπητέ φίλε, να σ' άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχει ε, άδικο αυτή τη φορά. Ξέρετε, δεν βλέπω αυτό το νόημα της, λέμε δηλαδή την προώθηση της καινοτομίας. Αλλά τελικά ε, προωθούμε τα λιγότερο καινοτόμα προβλήματα και κανένα αυτοκίνητο δεν θα απαγορευτεί. Απλά θα πρέπει να πληρώσω αν θέλετε ένα πρόστιμο. Τίποτα δεν πρόκειται να απαγορευτεί. αυτό. ευχαριστώ. Κυρία Βίλτς, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε στο θέμα αυτό. Έχουμε την ίδια αντιπαράθεση όπως αυτό των δυτικών δυτικής ρωσοχημάτων και γενικά τα θέματα που βλέπουμε στα αυτοκίνητα, ιδιωτικά ή επαγγελματικά, όλα αυτά χρόνια. Οι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν είναι αποδεκτές ακόμη και οι πιο μικρές ε, προϋποθέσεις ή περιορισμοί στην παραγωγή. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε σοβαρά προβλήματα ως προς εκπομπές των, ε, του διοξιδίου του άνθρακα ε, στον χώρο των μεταφορών. Πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και πρέπει και ο τομέας των μεταφορών να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων αυτών. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν με τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες και επεμβάσεις δεν προσέφερε έντιμο έργο και πιστεύω ότι είναι βέβαια αισιόδοξε οι τροπολογίε και ο κανονισμό με την αναθεώρηση μπορεί να βελτιώσει το κείμενο, μπορεί τα νομοθετήματα, αλλά δεν επαρκεί για να έχουμε προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα όρια εκπομπών για το 2020. Θα ήταν ε, ένδειξη αμελού συμπεριφορά, πιστεύω, εάν δεν προβλέπαμε πιο φιλόδοξου στόχου για το 2025. Φιλόδοξοι στόχοι λοιπόν και ανώτατα όρια που θα μπορούσαν για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να είναι ακόμη και ευνοϊκοί, να έχουν ευνοϊκή δηλαδή ε, συνέπεια γιατί ε, θα σήμεραν και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων. Οι μεγάλες δανειοδοτικές συμβάσεις βεβαίως και οι τράπεζες δεν δέχονται την απαγόρευση των συγκεκαλυμμένων επιδοτήσεων για τον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Κράμερ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βίλς ποιος μίλησε για προδιαγραφές και για προγραφές οι οποίες θα είναι αδύνατες να εφαρμοστούν από τι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, θα θέλετε να απαντήσετε, κυρία Βίλ. Ναι. Όλη η συζήτηση για τις ανώτατες ε, αξίες, για, τα, για τις τιμές είναι αδύνατη να εφαρμοστεί όταν αυτές οι αξίες δεν έχουν τεθεί πρώτα, όταν αυτές οι τιμές δεν έχουν οριστεί. Είμαι υπέρ πολύ αυστηρών ορίων για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία όμως να μπορεί να τηρήσει και πιστεύω ότι όσο περισσότερη πίεση ασκηθεί, πολιτική πίεση από τους κατασκε... Ε, προς τους εκατασκευαστές τόσο καλύτερη τεχνολογική Τεχνολογικέ εξελίξεις θα έχουμε και τόσο περισσότερα καύσιμα θα μπορούμε να ξεκονομήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την μπλε κάρτα την οποία <laughs> τραβήξατε μόλις τώρα, μάλιστα. Θα διαβάσω την λίστα των επόμενων ομιλητών, Πιλάρα Γιούζο, Κάρεν Φλόρενς και κύριο Μέρκινς. Κλείνει λοιπόν η λίστα των ομιλητών. Παρακαλώ. Κυρία Γιούζο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εδώ μιλάμε για μια βιομηχανία πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Μια βιομηχανία που έχει κάνει μια τιτάνια προσπάθεια με κόστος και προσπαθεί να εκπληρώσει τους στόχους της με καινοτομία. Μια λοιπόν βιομηχανία που συμπεριφέρεται καλά δεν κατανοώ γιατί πίεση για την πίεση. Ισορροπία, ναι, Προσοχή του περιβάλλοντος, αλλά όχι υπερβολική πίεση σε μια τόσο σημαντική βιομηχανία για την Ευρώπη. Έπειτα, με εκπλήσει το γεγονό ότι ένα κανονισμό που εγκρίθηκε το 2010 πρέπει να τροποποιηθεί τώρα. Και ξανά το 2014 λέτε. Ε, δεν είναι καλό αυτό και η μηχανή Η μηχανή χρειάζεται χρόνο για να μπορεί να προγραμματίσει τι επενδύσει, την καινοτομία κτλ. Οπότε με αλλαγέ καθε κάθε δύο-τρία χρόνια αυτό δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κράμα σε γενικέ γραμμές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να περιμένουμε τους νέους κύκλους δοκιμών που θα εναρμονιστούν σε εθνές επίπεδο για να μπορούμε να μιλήσουμε για στόχους πέρα από το 2020. Άρα ας μείνουμε στα 147 γραμμάρια που προβλέπονται για το 2020 και τελεία. Και μετά, αργότερα, θα έχουμε πιο πολλά επιχειρήματα, μπορούμε να δούμε τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα. Για να μπορεί να έχει χρόνο να ε, προγραμματίσει και η βιομηχανία. Για τα super credit συμφωνώ. Ε, για το 2016. Αρκεί να είναι το 50 γραμμάρια που είναι προς όφελος ε, των, των ηλεκτρικών οχημάτων και όχι και τα 75 γραμμάρια που καλύπτει και τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αυτά. Όχι άλλου στόχου γεμάτο το 2020 και διατήρηση των super credits. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φλόρεντς. Δεύτερος Κάλιστα, ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κάλαναν. Σε εκτιμώ, το ξέρεις. Βάλε για τα ακουστικά σου. Να σου κάνω και μία φιλοφρόνηση. Είσαι πολύ πιστός στη γραμμή σου, σταθερός, άκαμπτος. Και σήμερα το είδαμε αυτό. Επέμενες μέχρι τέλους. Πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπου η βιομηχανία είχε την άδεια να κάνει τα πάντα. Έχουμε γελιοποιηθεί, γελάνε μαζί μας. Έχουμε επιτρέψει τα πάντα. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γελάνε πίσω από την πλάτη των καταναλωτών. Να επιμείνουμε στους στόχους για το 2020 και θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε από τα παθήματα από την τελευταία συναδρία, ε, ε, συζήτηση πριν από ορισμένα χρόνια, τι ακούγαμε, θέλουμε χρόνο, θέλουμε χρόνο, δεν μας φτάνει, Χριστέ μου. Μάθαμε όμως από το πάθημα και τώρα πρέπει να βρούμε ένα διάδρομο για το τι θα γίνει μετά το 2020. Πιστεύω πως είμαστε πολύ χαλαροί και λυπάμαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήσασταν πολύ χαλαροί, δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει πολύ περισσότερα, να έχετε κάνει πολύ πιο θαραλές προτάσεις. Η αυτο, βιομηχανία μπορεί να κάνει αυτά που εσείς θεωρείτε συμβιβασμούς. Έχει τη δυνατότητα. Μην είστε τόσο ελαστικοί μαζί τους. Μην αγνοείτε, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους και είμαι τελείως κάθετος με, ε, με το επιχείρημα που λέω ότι τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, φιλελεύθεροι, ε, όταν θα τελειώσει η κρίση μας λέτε, τότε θα ασχοληθούμε. Όχι, τώρα, τώρα που βρισκόμαστε μέσα στην κρίση πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για το μέλλον. Τώρα, κύκλοι δοκιμών. Πραγματικά πιστεύω πως είναι γελία αυτή η συζήτηση. Θέλετε πραγματικά να παραμείνουμε εκεί που είμαστε. Πρέπει να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Κάθε μέρα στη Γερμανία κατασκευάζονται 10.000 αυτοκίνητα με λάθος προδιαγραφές, με λάθος τιμές. Ας μην επεκταθώ όμως αυτό. Πιστεύω ότι πραγματικά οι διαπραγματεύσει βρίσκονται σε σωστό στάδιο, ε, σωστό στάδιο. Θα οδηγηθούμε έργα και τώρα σε ένα συμβιβασμό. Τώρα, αν θα είναι 2015-2020, είναι άλλο πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τι εγγυήσει. Πραγματικά καταλάβετε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία τηρεί τα κατώτατα όρια εντάξει, ωραία, συμμερίζομαι τον πόνο σας, αλλά αυτά είναι πολι... πολιτικές απόψεις. Μάλιστα, yes we can, μπορούμε. Κύριε Μέρκης, κυρία Μέρκης μάλλον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω κι εγώ ε, στα όσα αναφέρθηκαν για τον κύκλο των δοκίμων. Για κοιτάξτε αυτήν την εφημερίδα όμως, θα, δείτε, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Πρώτη σελίδα. Απάτες στους, στις δοκιμές στα οχήματα. Και οι Βρυξέλλες επεμβαίνουν για να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό νομίζω ότι αρχίζει να το... Ε, για να εξηγήσουμε την κατάσταση, ο κύριος Γερμπράντη μάλιστα μιλάει στους δημοσιογράφους αυτής της εφημερίδας μας στο άρθρο, ε, είναι η κατάσταση αρκετά σοβαρή, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. γιατί ορίζεται ο κύκλος δοκιμής, αλλά μετά γίνονται κάποιες λοβιτούρες, γίνονται κάποιες ε, λαθροχειρίες, γίνονται κάποιε κάποιες μικροδιορθώσεις και τελικά δεν ε, υλοποιείται στην πραγματικότητα η δοκιμή αυτή. Οι φιλοδοξίε λοιπόν δεν είναι αρκετά φιλόδοξε και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα. Είναι απαραίτητο πια να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή αρχή. Δεν αρκούν 27 εθνικέ αρχέ ε, υπεύθυνε για αυτέ τι δοκιμέ. Τώρα, για τις πιστώσεις ε, είναι λάθος, είναι αντικίνητρο, δηλαδή ουσιαστικά ε, μπορεί να αποζημιώνουμε αυτόν που κάνει πιο πολύ καινοτομία, μεν, αλλά ταυτόχρονα, επειδή δεν είμαστε αρκετά αυστηροί, δεν ενθαρρύνουμε και τους άλλους ε, να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Καλό είναι να υπάρχουν αυτές τις πιστώσεις, αλλά, τα ανοίγματα πιστώσεων, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε και, εκείνους, και τους υπόλοιπους, αυτούς που δεν κινούνται χάρη σε μέγα ε, υπερ, μέγα πιστώσεις. Γιατί να μην ορίσουμε ένα σύστημα με θετικούς και αρνητικούς ε, πόντους, εφόσον κανείς ε, τηρεί πιο αυστηρούς κανόνες καινοτομίας, οι προδιαγραφές καινοτομίας, να ευνοείται περισσότερο με μεγάλες πιστώσεις, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε αυτούς που βρίσκονται στην πρωτοπορία και να σπρώχνουμε αυτούς που μένουν στα Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι ίσω να ήμασταν ε, φιλόδοξοι κάποτε, να θεωρούμασταν φιλόδοξοι, αλλά αν κοιτάξουμε άλλε περιοχέ του κόσμου, είναι πολλοί οι τομεί στου οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποτελεί ένα σημαντικό παράγωνα, το είπαμε και στο Δουβλίνο, ο κύριο Στάινερ, επικεφαλής του Διεθνού Προγράμματος για το Περιβάλλον, μίλησε για την έννοια της συνείδησης και την ε, ε, απώλεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Έννοια και τη πρωτοπορία αλλά και τη ανταγωνιστικότητα τη ε, βιομηχανία τη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, ε, χωρί βέβαια να γίνουμε υπερβολικά χαλαροί, να μην είμαστε και υπερβολικά απαιτητικοί στι προδιαγραφέ μα. Και τώρα θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το λόγο για να ακούσουμε μετά τον εισηγητή. Η Επιτροπή παρακαλώ. Φίλιπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κράμερ για την ε, συνοπτική παρουσίαση των τόσο πολλών τροπολογιών που και ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου που υπέβαλαν και τροπολογίε και εκείνα. Να ξεκινήσουμε με το στόχο των 147 γραμμαρίων για το 2020. Ο συνομοθέτη ζήτησε από την Κομισιόν να, να επιβεβαιώσει το κατά πόσον είναι επιτεύξιμο αυτό το στόχο. Αυτό κάναμε και μελέτη αντικτύπου καθιστά σαφέ ότι μπορούμε να τον επιτύχουμε με την διαθέσιμη τεχνολογία και με χαμηλότερο κόστο από ό,τι προβλέπαμε νωρίτερα. Όμως, εμείς δεν αποφασίσαμε ένα νέο τέτοιο αριθμητικό στόχο και λόγω περιορισμένης εντολής, αλλά και γιατί πρόσφατα υπάρχει μια συμφωνία και πρέπει να δοθεί α, βεβαιότητα στη βιομηχανία. Όταν τους δίνουμε ένα στόχο πρέπει να μείνουμε σε αυτόν. Ιδάλλως, πολύ ορθά και η βιομηχανία θα ήταν να αποφάσιμος. Και όπως και ο Σκράμερ πολύ ορθά λέει, και εσείς λέτε ότι α, θυμάμαι τις διαπραγματεύσεις που κάνατε κι εσείς για αυτό το ε, στόχο των 147 γραμμαρίων μέσα σε χιόνι στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, ε, μακροπρόθεσμα. Γνωρίζετε ότι και εμείς έχουμε πολλά έγγραφα πολιτικής όπως η Λευκή Βλώση για α, τις μεταφορές, για τον οδικό χάρτη, για ε, τη χαμηλή χρήση του άνθρακα και καταβάλουμε πολλές προσπάθειες για να μειώσουμε συνολικά την εκπομπή των ρήπων. Η Λευκή Βλώση για τις μεταφορές μιλάει για μείωση 120% στο 2030 των του ε, ε, και κατά 60% στο 2050. Αυτό αυτό λοιπόν για επιτευχθεί πρέπει να γίνει ενθέρωση τη νομοθεσία μόνο των δυνατών. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα και ασφάλεια για την βιομηχανία και για όλου του κοινωνικού ε, φορεί ώστε να ξεκάθαροι οι στόχοι. Αυτό όμως είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Οι μελλοντικοί στόχοι για να οριστούν απαιτούν βαθιά ανάλυση, εκτίμηση της διαθέσιμης μηχανής και, ε, τεχνολογίας και ποια θα είναι αυτή το 2025 για παράδειγμα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια έγκαιρη, ε, πρόορη ίσως αναθεώρηση ώστε να έρθουμε σύντομα σε εσά και προτείνοντα σας το προβλέψιμο μέλλον ένα νέο στόχο. Τώρα το θέμα των super credits. Εμείς δεν προτείναμε την ε, διατήρηση αυτού του καθεστώτος για πολλούς λόγους. Γιατί πρώτα απ' όλα κατανοούμε ότι τα υφιστάμενα που έχουμε ότι ο στόχος του 2017 των 175 ε, γραμμαρίων εύκολα μπορεί να επιτευχθεί και σήμερα. Άρα για ποιο λόγο να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για να μπουν τέτοια οχήματα στην αγορά, μάλλον οχήματα με χαμηλό ρήπο, όταν ήδη ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί σήμερα. Το Επίση, ο στόχο των αυτά 7 γραμμαριών μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλότερο κόστο. Οπότε, για ποιο λόγο να διατηρήσουμε τα σούπερ κρατήτη για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο δοκιμών, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κράμερ, ο οποίο λέει ότι αποφασιστεί για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να ισχύει και για τα εμπορικά οχήματα επίσης για τα επαγγελματικά ελαφρά οχήματα, γιατί ουσιαστικά είναι ε, παρόμοιε κατηγορίε, Οπότε πρέπει να υπάρχει συνέπεια και ακολουθία στην προσέγγιση. Κατανοώ όμω αυτό που λένε και οι γάμα, ε, συνάντηση στη ΓΔ δέλτα επιχειρήσεις, ότι είναι πολύ κοντά οι στόχοι και ειδικά η εισαγωγή του LTP στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και γι' αυτό λέμε κατάλληλη προθεσμία το 2017 για να εισαχθεί αυτό σε πλήρη εφαρμογή για τα γιοταχή και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Επ' αυτή την έννοια, αυτό που προτείνουμε τώρα είναι να προσαρμόσουμε τα αυθεντικά στοιχεία με την πρώτη ε, εισαγωγή του κύκλου δοκιμών αλλά πάντως σε πλήρη διαβούλευση με τη βιομηχανία, ώστε να μην είναι πιο αυστηροί κανόνας και να εφαρμόζονται ισότιμα στο μέλλον. Λοιπόν, κατανοούμε απόλυτα πόσο είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών και για αυτό το θέμα. Και το WLTP θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό στο μέλλον, θα δίνεται καλύτερη ενημέρωση στην κοινωνία στο μέλλον και αυτό θα ευνοεί καλύτερα τις μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιεί αυτά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Άλλε τροπολογίε επίση έχουν κατατεθεί, αλλά αναφέρθηκα στα θέματα κλειδιά, δηλαδή στόχοι, super credits και κυκλο δοκιμών και ευχαριστώ που δώσατε το λόγο να απαντήσω σε αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κράμερ, τα τελικά του σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ του αδέλφους που συμμετέχουν στη συζήτηση και κάνουν τι ε, παρατηρήσει του. Δεν θα επισέλθω σε αυτές που δεν έχουν σχέση με το θέμα μας, τη μεγάλη πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ και διάφορα σχήματα, αν θα πρέπει να είναι μεγάλα ή μικρά τα επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά είναι μια σημαντική μέρα σήμερα να το σημειώσουμε κύριε Ουν στο ημερολόγιο, διότι μπορώ να πω ότι προσυπογράφω όλα όσα ακούσαμε να λέτε. Σπάνια συμβαίνει αυτό, να συμφωνεί το Κοινοβούλιο με την Επιτροπή. Και θα ήθελα προ καταλαμβάνοντας αυτά που θα ακούσετε ενώ σχολιάζω, ε, να πω ότι προτίθεμαι να ετοιμάσω ένα κείμενο, ε, μια έκθεση την οποία θα ακολουθήσουν όλες οι προτάσεις και η οποία θα προχωρήσει απρόσκοπτα. Ξέρω ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές θέσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι δυνατό να το καταφέρουμε αυτό και αν όλοι δείξουμε μια κάποια κινητικότητα στα κύρια ζητήματα ε, που βρίσκονται επιτάπητος, θα τα καταφέρουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σας υποδείξω τις δικές μου προτεραιότητες που είναι σύμφωνες με, τον, με όσα είπε και ο κύριος Φιλπούν, ε, δεν πρέπει να ανατρέψουμε ή να παραβλάψουμε ή να αγγίξουμε το στόχο 2020. Βεβαίω θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε στι νέε συνθήκε, αλλά πρέπει να είμαστε και αρκετά δημοκρατικοί ώστε να ξέρουμε ότι μια συνενετική συζήτηση πριν από τρία χρόνια, η οποία θα πρεπει να μπορουμε να προσαρμοστουμε στις νεε πολλού συμβασμού, έστω και αν δεν ήταν όλοι σύμφωνοι, αλλά πάντω πέρασε από νομοθετική διαδικασία, σε μια κέρια σημασία ε, βιομηχανία όπως η αυτοκίνητο βιομηχανία πρέπει να εξασφαλίζει και ασφάλεια προγραμματισμού για, την, για τον κλάδο αυτόν. Άρα λοιπόν με έξι χρόνια μπροστά μας για το 2020 η αυτοκίνητο βιομηχανία χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο, ξέρετε, να προγραμματίσει την παραγωγή, το σχεδιασμό, ε, τα πρότυπα ότι είναι για τα ελαφρα, ελαφρα, ε, επαγγελματικά αυτοκίνητα πολύ περισσότερο από ότι για τα ε, επιβατικά. Άρα τα, τα σχέδιά τους για το 2020 και τα προγράμματά τους τα έχουν ήδη κάνει. Θα ήταν λοιπόν πολύ μεγάλο λάθος και μέσα σε περίοδο κρίση ιδιαίτερως να δώσουμε αυτό το μήνυμα, το κακό με εσφαλμένο μήνυμα ότι ανατρέπουμε πράγματα τα οποία θεωρούνταν εδρεωμένα. Το είπε και ο κύριος, και γι' αυτό θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καρσλούτερ, ότι Ασφαλώς και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την προσφορά ε, οικονομικών ε, οχημάτων για τον καταναλωτή. Δεν θέλουμε μεγαλύτερο κόστος, με πιο ε, αυστηρές προδιαγραφές για το 2020 όμως. Είναι αμφίβολο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Λίτσερ μπορεί να περιγράφει τον κόσμο όπως τον βλέπει, αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμος πάντα. Άρα λοιπόν μπορεί τα πράγματα να φαίνονται κάπω πιο δραματικά όταν τα περιγράφει εκείνο, αλλά υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τώρα, για το πώ θα είναι ο κόσμο μετά το 2020. Μπορούμε να κοιτάξουμε το κείμενο του κανονισμού. Ποιο είναι ο τίτλο του κανονισμού, Διατυπώσει εξασφάλιση των στόχων του 2020. Δεν είναι αυτό λοιπόν το κατάλληλο για να συζητήσουμε στόχους του 2025. Οτιδήποτε άλλο συζητούμε, είτε στους σκιώδες, είτε στις ομάδες εργασίας κτλ. Είναι ε, λόγια του αέρα. Και οι στόχοι που εξάπαντος πρέπει να τηρηθούν, και άλλωστε αναφέρθηκε αυτό και νωρίτερα, είναι οι στόχοι του 2020 και βέβαια χρειάζεται μία ε, μια μελέτη επιπτώσεων για την περίοδο μετά το 2020, γιατί μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση ως προς τα, επιβατικά, ως προς τα επαγγελματικά οχήματα κτλ. Μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλό να μην καταγράψουμε αριθμητικά στοιχεία μέσα στην έκθεση, τα οποία προδικάζουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακόμα κοιτάξει αρκετά προσεκτικά. Πάντως είμαι διατεθειμένος να κάνουμε συμβαστικέ ε, λύσεις, με προτεραιότητες όμως για μένα, την διαφύλαξη των στόχων του 2020, για όλα τα άλλα μπορώ να συζητήσω, εφόσον όμως καταλήγουμε σε υπεύθυνε και σοβαρέ λύσει. Συμφωνώ με στα υπόλοιπα με τον κύριο Φιλιππούν ότι μπορούμε ε, αντίθετα από ό,τι γίνεται στα επιβατικά αυτοκίνητα, να προωθήσουμε περισσότερο την ηλεκτροκινητικότητα στα επαγγελματικά οχήματα. Μετά υποδοθήκε από κάποιον άλλον συνάδελφο το ζήτημα της, ε, των κινήτρων ε, για την καινοτομία, γιατί αυτά τα οχήματα τα οποία έχουν πάνω από 50, 50 γραμμάρια εκπομπέ θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρικά οχήματα, να αντικατασταθούν δηλαδή από ηλεκτρικά. Εν πάση περιπτώσει, πάντα θα πρέπει να προωθούμε τη λύση των ηλεκτρικών. Ίσως μια κάποια αναφορά σε, σε μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να μπει στο κείμενο χωρίς να είμαι όμως δογματικά, δογματικός και απόλυτος στην υπόθεση αυτή. Αλλά πάντως ό,τι ορίσουμε θα πρέπει και να ε, υλοποιηθεί χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα εξουσιοδότηση ε, πράξαν και αυτό δεν είναι θέμα της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη πάντοτε ότι στο πλαίσιο αυτών των δύο νομοθετημάτων δεν, μπορούμε να, ε, δεν, δεν έχουμε να συζητήσουμε τις δοκιμές αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι υφίσταται αυτή τη στιγμή στην αγορά και το τι μπορεί να έρθει στο μέλλον. Αλλά πάντως βλέπουμε ότι αυτοί οι κύκλοι δοκιμών δεν προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και πρέπει ίσως να αναλογιστούμε ε, τι άλλο μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι και η αποδοχή αυτών των δοκιμών βλέπουμε να υποχωρεί σημαντικά, δεν είναι πιστή η καταγραφή των εκπομπών, δεν βοηθούν στον περιορισμό των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να επανεξεταστούν, αλλά δεν έχουν θέση στον δικό μας κανονισμό τώρα, ο οποίος έχει να κάνει με ε, την επιδίωξη των στόχων. Αυτά. Νομίζω. Παρακαλώ και τους και δυσηγητές να κοιτάξουν ε, λίγο περισσότερο τις λύσεις, μήπως μπορέσουμε να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις. Ήταν πολύ επικοδομητική στάση των πάντων και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε σύντομα να δούμε, να συζητήσουμε μια ε, δέσμη συμβαστικών προτάσεων για να καταλήξουμε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουμε σε 6 και 7 Μαΐου και στην Ολομέλεια θα εξετάσουμε το φάκελο τον Ιούλιο, κατά πάσα πιθανότητα. Μάλιστα, από τα ελευθερά επαγγελματικά οχήματα, λοιπόν, περνάμε στις ηλεκτρικές σκούπες. Εδώ ο Χόλγκερ Κράμερ έχει μία ένσταση. Και προτείνω, λοιπόν, να τον ακούσουμε από τα αυτοκίνητα στις σκούπες. Μάλιστα, είμαι 9 χρόνια εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο και έχω μιλήσει για πολλά τεχνικά και λεπτομερή ζητήματα και δεν ξέρω αν είναι λοιπόν σκόπιμο να μπούμε σε υπερβολικά τεχνικές λεπτομέρειες για έναν τέτοιον κανονισμό εφόσον είμαστε πολιτικοί. Δεν περίμενα να συζητήσω ένα τέτοιο θέμα για τις ηλεκτρικές κούπες εδώ πραγματικά. Και αυτό που θέλω να πω τώρα επί του περιεχομένου, ίσως να μην μπορείτε να το κατανοήσετε αμέσως. Έχετε στο μυαλό σας την ενεργειακή απόδοση. Τα τελευταία χρόνια, όταν χρησιμοποιεί κάποιος ηλεκτρική σκούπα στο σπίτι, αυτό έχει επιπτώσεις, δεν χρειάζεται. Πιστεύω πως δουλειά μας ως ευρωβουλευτές ως Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι να είμαστε πάρα πολύ κριτικοί απέναντι σε αυτήν την διαδικασία επιτροπολογίας, να την αξιολογήσουμε λεπτομερών και λεπτομερώς και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί αυτήν την απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Ε, δηλαδή, οι ηλεκτρικές κούπες πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικές. Έχουμε, κάνει πολύ, έχουμε πολύ καλές εμπειρίες από τα πλυντήρια και από άλλες οικιακές συσκευές Έχουμε δώσει δηλαδή πολύ καλές συμβουλές στους καταναλωτές ποια προϊόντα είναι ενεργειακά αποδοτικά, έχουμε τις ενεργειακές κλάσεις και όλα αυτά. Δεν αρκεί όμως. Δεν αρκεί όμως να τεθεί ο καταναλωτής ε, ρεύματος στο κέντρο, αλλά να δούμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε με ε, τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος του ίδιου. Πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι στην πολιτική μου καριέρα θα χρησιμοποιούσα αυτή την ε, φράση, αλλά η ικανότητα, η, προ... η... το δυναμικό τραβήγματος λειτουργίας της ηλεκτρικής κούπας είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να παραμερίσουμε. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ενέργεια, να δούμε τα, κιλοβάτ που χρησιμοποιούνται, που χρησιμοποιεί κάθε σκούπα στον οικολογικό σχεδιασμό. Υπάρχουν ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες που χρησιμοποιούν τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από άλλες, καθώς ανεβαίνει η, χρήση, καθώς αυξάνεται η χρήση, ανεβαίνει η κατηγορία. Δεν θα σας διαβάσω τα πάντα, αλλά τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία διατύπωσαν αμφιβολίες για τη διαδικασία της Επιτροπολίας, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία μεταξύ άλλων. Και θα το πω στα αγγλικά, γιατί το κείμενο είναι αγγλικό. Ε, λένε ότι το μήνυμα δεν είναι ξεκάθαρο για τον καταναλωτή. Οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες ε, μιλάνε για χρήση, για προτιμησιακή χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών ε, σκουπών, τα οποία Ενδεχομένως όμως έχουν υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας από ό,τι λένε. Πιστεύω ότι όσοι από εμάς προέρχονται από τη Γερμανία έχουν εμπειρία με μια πολύ καλή διαδικασία της ε, αρμόδιας ελεκτικής αρχής η οποία έχει διατυπώσει ότι το ισχύον ε, καθεστώς μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή, ε, πιθανές διακυμάνσεις, αποκλήσεις από όσα λέει τον χειρίδιο στον, ε, για την ενεργειακή κατανάλωση του κατασκευαστή και αυτό θα οδηγήσει στην ε, απώλεια εμπιστοσύνης του καταναλωτή στον ε, κατασκευαστή. Πραγματικά πρέπει να επεξεργαστούμε αυτές τις προδιαγραφές διότι Έχουμε μια οικολογική ατζέντα, έχουμε μια φιλική προς το περιβάλλον ατζέντα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς προς αυτή. Δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς διαφορετικά. Δεν θα εμπιστεύονται ούτε καταναλωτές τους κατασκευαστές, ούτε καταναλωτές εμάς τους πολιτικούς που δημιουργούμε τις προδιαγραφές για τους κατασκευαστές. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να κοιτάξουμε πραγματικά τις προδιαγραφές για τις ηλεκτρικές σκούπες και τη λειτουργία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μια ηλεκτρική σκούπα πρέπει να λειτουργεί και τελειώς μαζεύεται σκόνη, κύριε Κράμερ. Εντάξει, τώρα η διατύπωση ε, υπόκειται σε εσά. Εντάξει, είναι κάτι που σας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, είναι κάτι που προκαλεί αντιδράσεις, έχουν ήδη ζητήσει το λόγο συνάδελφοι. Πέτερ Λίζε, Κριστέιβι, Σοφή Οκουνή και η Λίντα Μακέβαν και ο κύριος Γκερμπράντι. Μήπως θα έπρεπε να διαβάσω αυτούς που δεν έχουν ζητήσει να μιλήσουν για τις ηλεκτρικές σκούπες. Φρέντερικ, είσαι πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θυμάμαι χρόνια πριν που ζητούσαμε αυτή την οδηγία για τον οικολογικό συνδυασμό 2005, αν θυμάμαι καλά. Δουλέψαμε πάρα πολύ το θέμα αυτό και ο Πίτερ ήταν εδώ και το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι και τις συζητήσεις με την Επιτροπή. Να μην ξεχνάμε τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει τότε και που παραμένουν και σημερινές προτεραιότητες, δηλαδή να έχει ελαχιστοποιηθεί το, στο μότο δυνατόν ο αρνητικός δίκτυπος για το περιβάλλον, ε, σε μία σειρά προϊόντων ενεργοβόρων και αυτό αφορά από το στάδιο της κατασκευής και σε όλες τις φάσεις του βίου του προϊόντος έως το τέλος του κύκλου ζωής. Κατανοώ αυτό που επισημαίνει ο κύριος Κράμερ. Εγώ δεν το αμφισβητώ. Βάσει του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου ε, υπάρχει αυτό το δικαίωμα το θέμα που τίθεται όμω εδώ είναι το εξή, γιατί διάβασα την ένσταση του κ. Κράμερ και κυρίω του λόγου των ε, αντιρρήσεών του και συμφωνώ με την ε, τοποθέτησή του προ την ε, ουσία που είναι ένα πρακτικό ζήτημα, αλλά από την άλλη τον μιλάει για την διάγνωση, για τους, ε, για τις ηλεκτρικές σκούπες που δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώς ε, ε, την απόδοση των ηλεκτρικών σκουπών που αναφέρεται σε έναν μαθηματικό, φυσικό τύπο που βρίσκεται στη σελίδα 11 της μελέτης και έχω κάνει πολλές μελέτες και υπολογισμούς, μαθηματικούς αλγορίθμους και όλα αυτά σε μια άλλη ζωή, αλλά όπως είπε και δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Από την άλλη νομίζω ότι έχω εκλεγεί από το ψηφοφόρο για να ακούω και τους ειδικούς τους ειδικούς της Επιτροπής που είναι ε, αυτή η δουλειά τους που πέντε χρόνια τώρα ασχολούνται με τα, με εφαρμοστικά αυτά μέτρα της οδηγίας ε, οικολογικού σχεδιασμού αλλά και όλους τους εμπειρογνώμενους εμπλεκόμενους φορείς, την ε, βιομηχανία κτλ που σχεδόν ομόφωνα πλην ορισμένων και διγερμανών συμφωνούν, υποστηρίζουν την πρόταση αυτή όπως έχει διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία προβλέπει νομίζω γιατί είναι και αυτό μία περίοδο σταδιακής εισαγωγής. Δεν ε, προβλέπεται παρά μόνο ε, κάποια χρόνια μετά να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτή για, για τη βιομηχανία. Άρα, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, γιατί εδώ ε, αυτό έχει να κάνει με, το μαθηματικό ε, τύπο, άρα η επίδοση της ε, συλλογής των, ε, της σκόνης προβλέπεται, στο, περιλαμβάνεται στον τύπο ο εισηγητή λέει όχι, όλοι οι άλλοι όμω λένε ναι και εγώ τίνω να συμφωνήσω με την πλειοψηφία και άρα υποστήριζω την πρόταση επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι που έχουμε την ευκαιρία να τα συζητούμε όλα αυτά με διαφανή τρόπο τώρα, αλλά θα πρέπει και να είναι σαφές ότι πλην μίας όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ε, που αφορά αυτή η ε, πρόταση τη θεωρούν θετική Έχω λάβει πολλές ε, επιστολέ από επιχειρήσει που αρχικά ήταν επιφυλακτικέ, αλλά τώρα την ε, υποστηρίζουν την πρόταση, γιατί έχετε μεταξύ Έχω δει κράτη-μέλη τα οποία ήταν επιφυλακτικά, όπω το Βέλιο και η Γερμανία αρχικά, και που εν τέλει, από ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον ύστερα διαπραγματεύσει και τι συζητήσει έχουν συμφωνήσει στην ε, οδηγία Eco Design η ουσία είναι ότι προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και πόρους, πράγμα το οποίο δεν είναι στην, στη λεπτομέρειά του, στην εφαρμογή του, τη λεπτομερή απλή υπόθεση, αλλά πάντως αποτελεί ένα θετικό μέσο, ένα καλό εργαλείο και πολλές είναι οι επιστολές που βλέπουμε και που λένε ότι εν τέλει συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις. Έχω συστήσει επιμακρών με τους ειδικού και ιδιαίτερα με την ε, με τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, μας ενθαρρύνουν ε, και θέλουν να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, από τη Βεσφαλία, τη δική μου εκλογική περιφέρεια ιδιαιτέρως. Και... Ε, από την Επιτροπή, από διάφορες επιχειρήσεις που έχω συζητήσει και από διάφορους εμπλεκόμενους βλέπω ότι, όπως είπε και η κυρία Φρεντερικ ΡΙΣ θα πρέπει να υποστηρίξουμε την... ε, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση του συναδέλφου. Τώρα στο συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω από την αίθουσα, έχω ένα άλλο θέμα για να συζητήσω. Ε, πάντως ευχαριστώ ε, και θα ήθελα να πω ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρώτον, και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί είναι καλή και χρήσιμη αυτή η πρόταση Εντάξει, συμβασμός, ε, ο μόνος τον οποίο κατέληξε η πλειοψηφία, γιατί διαφορετικά δεν θα εξασφαλιζόταν κτλ. Ε, διότι ε, η κυρία Λάτσινγκ το είπε, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω για όλους, πριν ψηφίσουμε, ότι αυτή είναι μία, λύση, μία θέση. Και δεύτερον, η εμπλεκόμενη επιχείρηση, οι επιχειρήσει οι οποίε υποστηρίζουν την πρόταση λένε ότι με την τροποποίηση του τύπου μπορεί να φέρνουν αποτελέσματα. Πάντως ε, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν αυτά τα επιχειρήματα, ώστε να γνωρίζουν όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν ε, ποια είναι τα δεδομένα. Ευχαριστώ, Chris Davis. Πρόεδρε, είπατε στο παρελθόν ότι θέλετε αυτή η επιτροπή να, γίνει, να έρθει πιο κοντά στο κοινό και συμμερίζομαι ε, το είπα και στην ομάδα μου χθε. Ε, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να φέρουμε τις δικές μας ηλεκτρικές κούπε και να κάνουμε και ένα flash dance με αυτές και χορογραφίες. Ωστόσο, σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Δύο μάλλον σύντομέ ερωτήσει. πόσοι κατασκευαστές έχουν φέρει αντιρρήσει σε εσά συγκεκριμένα, στι προτάσει σας, πόσε εταιρείε. και Εάν αλλάζετε αυτή την πρόταση, αλλάζετε τη διατύπωση, την εξισορροπούσατε κάπως ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό θα οδηγούσε σε κλονισμό της ισορροπίας, θα είχαν άλλες εταιρείε παράπονα για άλλους λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Chris Davis, Σοφή Οκουνή, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δική μου παρέμβαση έχει να κάνει με την ρώτηση του κυρίου Λίσε προς την Επιτροπή, δηλαδή το να εξετάσουμε ακριβώς γιατί αυτό το κείμενο και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο. Ωστόσο δεν ήθελα εγώ να πω το εξή, γιατί λυπούμε πολύ που είμαι υποχρεωμένη σήμερα να πω στους ε, συμπολίτες μου στην Ευρωπαϊκή Εκλογική Περιφέρεια ότι έχω να συζητάω Προδιαγραφέ για σκούπε ηλεκτρικέ. Δεν έχουμε τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε να κάνουμε. Ζούμε μια συγκυριακή κρίση που είναι οικονομική, δημοσιονομική, κοινωνική, δημόσια υγείας, περιβαλλοντική. Ζούμε δυσκολίες σε κάθε πεδίο και σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Δεν θα έπρεπε να έχουμε άλλες προτεραιότητες από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα να συστήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορούσε να αφήσει κατά μέρο τέτοιου τύπου εκθέσεις οι οποίες, ας τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα, είναι θέματα λεπτομέρειας και να τα συγκρίνουμε με την προηγούμενη σύνοδο, την απόρριψη του backloading των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, της οπισθοβαρούς μέτρησης, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία και την ε, ποιότητα του κρέατος. Γιατί δεν μπορούμε να τους προστατέψουμε κύριε Πρόεδρε τους πολίτες όταν έρχεται ένας απατεώνας και εμφυτεύει... Ε, εμφυτεύματα στήθους με συνθήκες παραγωγής απαράδεκτες που ε, καταστρέφουν τη ζωή και την υγεία τόσων πολιτών της Ευρώπης, κατοντάδων και περισσότερων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια μείζωνα οικονομική κρίση, εμείς, η Επιτροπή του Περιβάλλοντος και ο Καλχάιντς Φλόρεντς το είπε πολύ καλά προηγουμένως, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτά τα οποία ζούμε σήμερα και η οποία είναι, ε, εντάσσεται μέσα σε μια έκφραση που μπορούσε να ακουστεί ως θεωρία ε, ότι περνάμε από την κρίση και από την καταστροφή πριν περάσουμε στα καλύτερα. Ναι, αλλά πρέπει να, λήξει, να αλλάξει βιομηχανικός κύκλος ε, νέα, ε, νέα νέες λύσεις, ε, νέες προτάσεις αστικές. Αλλά ας αφήσουμε τις κούπες για όταν τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα κύριε Πρόεδρε. Ναι, το καλύτερο θα ήταν η σκούπα να λειτουργεί με ανανεώσιμη ενέργεια. Δεν θα είχαμε λοιπόν τότε τόσα πολλά λεπτά σωματίδια σκόνης. Επόμενο συνάδελφος. Ε, ε, πρέπει να σας πω βέβαια αγαπητοί συνάδελφοι ότι όταν ε, είναι έργο μας ως κοινοβούλιο πρέπει να τα συζητάμε όλα, πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα στα σοβαρά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι κι αλλιώς. και ο συνάδελφο, πρέπει να πάρει μόνιμη η θέση εδώ πέρα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρία επιτροπών συζητήσαμε και ήταν πάλι εδώ και πιστεύω πως είναι ε, σημαντικό αυτό. Έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία από τη μία ε, είναι συγκεκριμένα και πρέπει να τα ενισχύσουμε και πρέπει να, θέσουμε, να έχουμε ε, συνολική θέση των πραγμάτων, να μπορούμε να αιτιολογήσουμε, να μπορούμε να δώσουμε το background, να πούμε γιατί ναι ή γιατί όχι. Τώρα ναι, ξέρω ότι, από το, ε, ότι το, το να συζητάμε σκούπες αντί για backloading φαίνεται κάπως παράξενο. Τέλος πάντων, επόμενη ομιλήτρια, κυρία Λίντα Μακέβαν. Συμφωνώ, Πρόεδρε, μαζί σα. Παλέψαμε τόσο πολύ να αποκτήσουμε αυτές τις εξουσίες, να έχουμε λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και εντάξει, μπορεί να λέμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά Θυμάστε εκείνη την πρόταση που καταφέραμε να μπλοκάρουμε να μπει μια τόσο τοξική ουσία στο κρέας. Λοιπόν, ε, ε, ναι, μπορεί να μην φαίνονται εκ σημαντικά τα ζητήματα, αλλά είναι και αυτό είναι σημαντικό θέμα γιατί αφορά την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και όπω είπε ο Chris Davis, ε, πράγματι θυμάμαστε πώς διαφωνούμε και πώ συμφωνούν με την πρόταση Κομισιόν. Και θυμάμαι τι μα είχε πει η Κομισιόν τότε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπήρξε διαβούλευση με τι επιχειρήσει και φαίνεται ότι επελήθη το πρόβλημα ουσιαστικά εκτό από μια εταιρεία. Άρα η Κομισιόν έκανε τη δουλειά τη ουσιαστικά και δεν μπορεί η ομάδα μου να υποστηρίξει τον κύριο Κράμαρ. Δεν υπερεύει ε, τις που έχει η Κομισιόν, οπότε δεν θα την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα Μακέβαν. Κύριος Γκυρμπράντη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους προλελήσαντες, όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κράμερ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο προσπάθησε, ασχολήθηκε με το θέμα, δέκα διαφορετικές ηλεκτρικές σκούπες, κοίταξε για να δει λοιπόν ποιος είναι, ποια ήταν η καλύτερη, ποια έχει την καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης και πραγματικά Αυτό ήταν και αυτό που, θα, που είχε ζητήσει και το Συμβούλιο από την Κομισιόν, δηλαδή να ασχοληθεί εντελεχώς, να εξετάσει εντελεχώς το ζήτημα έτσι ώστε να κάνει μια περιστατωμένη πρόταση. Κύριε Πρόεδρε όμως, Μπορούμε να διεξάγουμε μια τέτοια συζήτηση, σίγουρα. Αυτό που φοβάμαι όμως είναι ότι μπαίνουμε τώρα στα, σε μια συζήτηση για οδηγία, για σχεδιασμό και ρίχνουμε ενδεχομένως αλάτι στις πληγές. Πρέπει να είμαστε παρόντες ενώ συντελούνται αυτές οι αλλαγές. Πρέπει να είμαστε παρόντες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ε, αλλαγή, ένα βιώσιμο νέο σχεδιασμό και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Εδώ πέρα βλέπετε, μειώνεται ο πάγος στη, στη Γρυλανδία. Λιώνουν τα παγόβουνα, πρέπει να σκεφτούμε βιώσιμα. Και όλα σχετίζονται με αυτό. Το πρόβλημα της αρχικής πρότασης ήταν ότι το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να ασχοληθεί με το πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα, έτσι όπως είναι, δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν λυμένο. Πρόεδρε, μόνο για να απαντήσω στα όσα είπε η κυρία Οκονή, συνάδελφο, δεν θα κάνω τη συνήγορα τη Επιτροπή, δεν το χρειάζεται καν, αλλά και ξέρω ότι μερικέ φορέ στο Παρίσι αρέσκεται να ε, βάζει το δόλιο του κατηγορουμένου την Επιτροπή, αλλά ε, κοιτάξτε, δεν είναι εδώ η Επιτροπή η οποία φέρνει την υπόθεση για συζήτηση. Η, ένσταση είναι αυτή που φέρνει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μέτρα εφαρμοστικά, τα οποία έχουν προσδοριστεί από μια οδηγία ε, του οικολογικού σχεδιασμού, που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο και εργαλείο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να μιλάμε λοιπόν για σκούπες ηλεκτρικές και για μαθηματικούς τύπους, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σημαντικό. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Κράμερ. Ναι, δεν θέλω να καθυστερήσω τώρα, αλλά ένα πράγμα θέλω να επισημάνω για να απαντήσω σε κάτι το πολύ σημαντικό. Ότι στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουμε, είτε πρόκειται για τα ελαφρά επιβατικά που συζητήσαμε, είτε που έχουν επιπτώσει στην βιομηχανία από την νομοθεσία μα. Πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα τη βιομηχανία. Λοιπόν- Τώρα, λοιπόν γιατί αλλάζουμε στάση. Βεβαίω οι επιχειρήσεις οι οποίες... Χρειαζόμαστε προϊόντα τα οποία Χρειάζονται νέες επισημάνσεις. Το θέμα δεν είναι να πάρει το προϊόν την ε, καλύτερη επισήμανση. Το θέμα είναι να πληρεί τις προδιαγραφέ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι οι μηχανές της BOS τα μηχανήματα της Bosch και της ε, Siemens από το Φεβρουάριο του 2013, πριν από δύο μήνες δηλαδή, η εταιρεία αυτή διατύπωσε τις εντονότατες ανησυχίες της ε, για την, για την αναδιατύπωση τις οδηγίες για τις ηλεκτρικές σκούπες. Εντονότατες λοιπόν ανησυχίες. Και από τότε μέχρι τώρα δεν έγινε καμία αλλαγή στη διαδικασία επιτροπολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα ποιε εταιρείε είναι αυτέ που υποστηρίζουν την αλλαγή στι ε, ηλεκτρικέ σκούπε. Εγώ λέω δεν πρέπει να ρωτάμε τις ίδιες εταιρείε τι πιστεύουν. Όχι, να δώσουμε το θέμα σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διότι διαφορετικά έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, έχουμε επέμβαση της βιομηχανίας στην νομοθεσία. Μάλιστα. Ο πρόεδρος. Βλέπω εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά βλέπω ότι κάποιοι μιλάνε αλλά πραγματικά, ναι, όντω υπάρχουν, συμφέροντα, υπάρχουν ορισμένοι που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπό τη, για να μα ενημερώσει για το πού βρισκόμαστε σχετικά με τι ηλεκτρικέ κούπε, τι έχουν δείξει οι δοκιμέ, ποια τα αποτελέσματα των μελετών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία που μας δίνετε να πάρουμε και εμείς το λόγο. Είναι κομμάτι του δημοκρατικού διαλόγου να κάνουμε αυτή τη ζήτηση, να ακούσουμε τις σοβαρές συνστάσεις, αν υπάρχουν, τις οποίες πάντα λαμβάνουμε σοβαρά. Κύριε Χωνή, να πω ότι Φυσικά και δεν είναι τόσο σημαντικό στο backloading όπως και πολλά άλλα θέματα, αλλά συλλογικά η ενεργειακή απόδοση είναι πολύ σημαντικό θέμα και πώς μπορεί να επιτευχθεί η ενεργειακή απόδοση με τόσες μικρές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει ισοδύναμο για να βάλουμε μια άλλη υποχρέωση γενικά στο ηλεκτρικό ε, κλάδο, πρέπει να μπει στις λεπτομέρειες. Και μόνο αντί στις λεπτομέρειες ε, μπορείς να επιτύχεις το στόχο. Τώρα για αυτή την πρόταση, με αυτό τον, θα κερδίσουμε 19 ε, τεραργατόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όπως ε, οι καυστήρες νερού, αλλά σίγουρα θα εξοικονομήσουμε χρήματα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Θα είναι πολύ σημαντικά τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και ήταν ε, κεντρικό στοιχείο συζήτηση που είχαμε με τα ενδιαφέρομενα μέρη και στη διαβούλευση ε, και στην ε, Κανονιστική Επιτροπή ήταν πάντοτε ε, κεντρικό θέμα αυτή η πρόταση. Η απόφαση της Κανονιστικής Επιτροπής ήρθε με συμβασμό μόνο αν εκρατός μέλος δεν ήθελε να δεχτεί αυτό το συμβασμό. Τουλάχιστον η Κανονιστική Επιτροπή κατέληξε μια θέση που μπορούμε να προωθήσουμε. Μια θεμητή ανησυχία που εκφράζεται. Γιατί όταν βάζουμε την ετικέτα αποδοτικότητας στις ηλεκτρικές σκούπες α έως g, μπορεί να έχεις μια σκούπα που να έχει α στην αποδοτικότητα, αλλά τελικά να κάνει πολύ κακά τη δουλειά καθαριότητα. Δεν υπάρχει σήμερα, αλλά ουσιαστικά μπορεί να συμβεί. Μπορεί να έχουμε ένα κακό προϊόν και με αυτό που κάνουμε, με αυτή την νομοθεσία, μπορεί να έχουμε στράγγλωση τη αγορά. Αυτό που προσπαθήσαμε να λύσουμε κάνοντας μια αλλαγή ε, που προτείναμε στην Κανονιστική Επιτροπή, απαγορεύοντας αυτό τον τύπο ηλεκτρικών ε, σκουπών. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπετε εσείς μπροστά σας διαφέρει από την αρχική πρώτη Κομισιόν ακριβώς γιατί προβλέπει απαγόρευση για τέτοιου είδους ε, ανεπιθύμητα προϊόντα τη μέρα που θα τεθεί η ισχύ νομοθεσία περί ετικέτας. Άρα, κατά τη γνώμη μας, ε, διασκεδάζεται αυτή η ανησυχία με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, αλλάζονταν περαιτέρω λεπτομέρειε στην εξίσωση με την οποία υπολογίζουμε την ενεργειακή απόδοση. Ούτε να πολλαπλασιάσουμε επί δυόμιση ε, το βάρο που δίνουμε σε αυτή την εξίσωση ε, για το πόσο καλή είναι η ηλεκτρική σκούπα στην ισχύ απορρόφησης τη κόρνη από το πάτωμα και τα χαλιά. Αν αντίθετα το κάνουμε αυτό, αυτό θα αντίκειται στην τεχνική και επιστημονική βάση που ακολουθούμε και είναι πολύ σημαντική για να γίνεται αυτή η εκτίμηση. Ο αριθμό που βλέπετε στην πρώτη είναι 0,2 και σα ζητούμε να δεχτείτε την αλλαγή του 0,5. Πηγαίνοντας στην Εκανονιστική Επιτροπή είχαμε προτείνει 0,15 γιατί είχαμε δύο αποδείξεις από τη δική μας προπαρασκευιστική μελέτη και μία από την Πορ Siemens που υποστήριζαν τον βιορυθμό. Όμως οι βελικές αρχές έκαναν ε, τις δικές τους δοκιμές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 0,2, μια ψηρότερη δηλαδή τιμή, ήταν πλέον κατάλληλη. Εξετάσαμε λοιπόν προσεκτικά και την πολύ καλή δουλειά που έκανε οι αρχέ. Είδαμε και τα τρία στοιχεία από εκείνο και έτσι τροποποιήσαμε το 0,15 σε 0,2. Θεμητή αλλαγή, μια αλλαγή που κινεί στη κατεύθυνση και δεν υπάρχει καμία βάση που μας απαγορεύει να πάμε με το 0,15 στο 0,2, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο 0,5. Και ελπίζω να σας απαντώ κύριε Λίζε. Φοβούμαι ότι αυτό θα είναι πολύ ε, επικίνδυνο βήμα. Δηλαδή να εισάγουμε μία τιμή που δεν έχει καμία επιστημονική βάση και είναι τόσο μακριά και από την ε, βελγική μελέτη. Για να απαντήσω στον κύριο Ντέιβις, ο οποίος έστειλε τον αριθμό των επιχειρήσεων που βλέπουμε αρέσει και την πρόταση. Πριν πάμε στην Κοινωνική Επιτροπή, δύο εταιρείε εξέφρασαν ανησυχία για αυτό το ζήτημα και από την υιοθέτηση των αλλαγών από την Επιτροπή, λαμβάνοντα υπόψη τι πληροφορίε που λάβαμε, μόνο μία είναι επιχείρηση που συνεχίζει να εκφράζει δυσαρέσκεια με την κατάσταση. Επίσης να προσθέσω ότι αν κάναμε αυτή την αλλαγή στην πρόταση οικολογικού σχεδιασμού, θα έπρεπε να κάνουμε αντίστοιχη αλλαγή και στην πρόταση για την ετικετοθεσία, γιατί είναι ήδη μεθοδολογία για τις δύο προτάσεις. Άρα θα παραλαμβανούσαμε τον ε, καταναλωτή γιατί θα του δίναμε μία εξίσωση για να κατανοεί την σχετική απόδοση της ηλεκτρικής κούπας χωρίς να είναι η ευθύ εξίσωση. Δεν θα το κάναμε αυτό με κανέναν ε, με καμία χαρά. Λοιπόν, ε, δεν αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε αυτό το ψήφισμα, αλλά δηλαδή την πίεση που ασκεί γενικότερα το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή σα, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε ό,τι εκκρεμεί από το eco-design, γιατί αισθανόμαστε άσχημα, γιατί σας προσχεθήκαμε μία σειρά πραγμάτων και καθυστερούμε. Τώρα προσπαθούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφο. σημαίνει ότι θα κάνουμε πιο σύγχρονε συζητήσει. συζητήσεις, θέλουμε τι συζητήσεις και αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι συζητήσει να είναι επικοδομητικέ, ώστε και εμεί σα πληροφορούμε όσο γίνεται πιο συστηματικά. Είμαστε ανοιχτοί γι' αυτό και περιμένω να ξανάρθω για την ίδια συζήτηση στην Επιτροπή σας και στο μέλλον. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση πρόσθετη. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην συζήτηση. Και πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Το σημείο 10. Με συγχωρείτε κύριε 8. Η δική μου έκθεση. Μάλιστα. Ακριβώς λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο μόλις συζητήσαμε και πιστεύω ότι είναι ναι, ένα θέμα το οποίο δεν συζητούμε όσο θα έπρεπε. Οι πράξεις καταξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, τις ε, διαπραγματεύσεις το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά στον τριμερή διάλογο, ότι στο τέλος όλα καταλήγουν στις πράξεις εξουσιοδότηση ή στις εκτελεστικές πράξεις και πιστεύω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε αρκετά γενναιόδοροι ενδεχομένως. Μάλιστα. Δεν ήθελα να ενοχλήσω τη συνάδελφο από το τηλεφώνημά της, ήταν σημαντικό φαίνεται. Θέλαμε λοιπόν, όπως έλεγα, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχει έρθει η ώρα να το α, να λύσουμε. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση που θα καταρτήσει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και εμείς έχουμε ζητηθεί να γνωμοδοτήσουμε. Μπορούμε, πιστεύω, να υποστηρίξουμε απόλυτα την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ως Επιτροπή Περιβάλλοντος και ως ε, εισηγητής συνέταξα μια γνωμοδότηση την οποία θα μεταβιβάσω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και θα σας την παρουσιάσω πολύ συνοπτικά. Εμείς μόλις είδαμε, μόλις τώρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, ζητήματα. Πολλές φορές είναι και ευτελή, ξέρω εγώ, ικανότητα απορρόφησης μιας ηλεκτρικής κούπας. Μόλις, μόλις το είδατε. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία ε, είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα των πρόσθετων τροφίμων, οι δραστικές ουσίες, η επισήμανση των τροφίμων, ε, εισαγωγές από την ε, Ιαπωνία, τροφίμων από την Ιαπωνία. Πάρα, πάρα πολλά πράγματα αφορά όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ζήτημα αυτό σήμερα φάνηκε ξεκάθαρα η θέση των πολιτικών ομάδων ε, όταν συζητήσαμε για τις σκούπες. Πιστεύω όμως ότι είναι δουλειά μας, είναι αρμοδιότητά μας να θέτουμε αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να τα ελέγχουμε, διότι αυτός είναι και ο ρόλος μας και όλας διεξαγωγή ελέγχου. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα της έκθεσης. Πολιτικές αποφάσεις, λήψη πολιτικών αποφάσεων. Πολλά από αυτές, ε, πολλά από αυτές ζητήματα για τα οποία προτείνει Παράξη κατά εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις η Επιτροπή είναι πολιτικά ζητήματα και όχι μόνο τεχνικά. Τι σημαίνουν οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση, να σας ρωτήσω, ξέρετε. Μήπω πρέπει να κάνουμε ένα σεμινάριο επιμορφωτικό από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και μετά. Έχουμε αναλάβει πρόσθετε αρμοδιότητε και πρέπει να τι λάβουμε σοβαρά υπόψη και να τι ασκήσουμε. Και πολλέ φορέ έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι το τα προσπερνάει όλα αυτά. Εμεί, λοιπόν, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε συντάξει μια τέτοια, ε, αυτή είναι εδώ τη γνωμοδότηση, διότι είναι απαραίτητη. Είναι, υπόκειται απόλυτα στι αρμοδιότητέ μα. Τώρα, έχει, έχουμε ένα λεπτό. Έχει μια συνάδελφος ζητήσει το λόγο, η εισηγήτρια στην νομοδότησή μου και... Όχι, δεν θέλετε να μιλήσετε, τότε ο Chris Davis, ο επόμενο ομιλητής. Μάλιστα, θα είμαι σύντομος. Υποστηρίζω τα σχόλιά σα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι συνεχιζόμενο. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Πιστεύω ότι πέραν του ψηφίσματος που έχουμε εδώ, ε, δεν γνωρίζω τι συζητήσεις διεξάγονται αυτή τη στιγμή για το πώς ε, πρέπει να συνεχίσουμε, αν θα... Αν έχει γίνει οποιαδήποτε συζήτηση σε οποιαδήποτε επίπεδο, ή προεδρικό, είτε και χαμηλότερο, για να συζητήσουμε αυτές τις ε, λεπτομέρειες. Σίγουρα μπορούν να συνεισφέρουν και οι άλλες επιτροπές. Έχουν μάλιστα παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο έχει διατυπώσει την ε, αντίρρησή του και εμείς ως Κοινοβούλιο καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε αυτές τις αντιρρήσεις. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε επιτροπή-επιτροπή, λιθαράκι-λιθαράκι. Να δούμε στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε πετύχει να ξεπεράσουμε τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου στις περιπτώσεις που έχουμε καταφέρει να, να ξεσκεπάσουμε ως ε, αδύναμη την ε, θέση της Επιτροπής του Συμβουλίου, είχαμε να σας πω και ένα παρόμοιο θέμα στην Επιτροπή Αλληλείας. Βέβαια, κράτησε πάρα πολύ καιρό, αλλά αυτό γιατί συνέβη. Αυτό συνέβη γιατί και η Επιτροπή και το Συμβούλιο αρνήθηκαν να καθίσουν και να συζητήσουν μαζί μας. Αρνήθηκαν να καθίσουν και να βρουν λύση ρεαλιστική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να σε έκανε άλλο στο... Α, κύριε... Κύριε Χάση. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. Τις προτάσεις του Chris Ντέιβις τις θεωρώ πολύ χρήσιμες. Όλοι τουλάχιστον όσοι έχουν συμμετάσχει στους τριπερίες διαλόγους ξέρουν πως πάντοτε το Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για να ε, καταφέρει να περάσουν εκτελεστικές και όχι κατευθυντώτες πράξεις. Και χθε ήμουν μια τέτοια συνάντηση, όπου συζητούνται κανονιστικές διαδικασίε με έλεγχο βάσει προηγούμενης ε, προηγούμενου καθεστώτος πέντε τέτοιες διαδικασίες έγιναν εκτελεστικές πράξεις. Αν και τα κριτήρια στην παλιά συνθήκη σχετικά με την καπνιστική διαδικασία με έλεγχο είναι ίδια με τα κριτήρια που ισχύουν τώρα για την επιλογή πράξεων κατοξιοδότηση και επ' αυτού θα ήθελα να είμαστε πιο δυνατοί, πιο συγκεκριμένοι και θα ήθελα πιο ισχυρή διατύπωση από τον Ματία στο κείμενο για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα συμφωνώ κι εγώ Ακούγεται πάρα πολύ βαρετό αυτό το θέμα. Πόσο συναρπαστικό μπορεί να το βρει κανείς, αλλά είναι σημαντικό. Αυτά ευχαριστώ. Ναι, τώρα δεν βλέπω άλλο να ζητάει το λόγο. Και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή καλωσορίζει τη συζήτηση του θέματο αυτού στο Κοινοβούλιο. Είναι καλή η ευκαιρία καλός ο χρονισμός και η εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα. Βεβαίω, μπορεί κανεί να πει ότι λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα, γιατί ήδη έχουμε υιοθετήσει περί τη 55 κατεξουσιοδότηση εν Απρόσκοπτα δουλεύει σχετικά. Συνηθίζουν νομίζω και τα όργανα να αξιοποιούν αυτό το νέο σύστημα. Βέβαια υπάρχουν πολλές συγκρούσεις στις νομοθετικές διαδικασίες και ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό των ορίων. Εδώ δεν έχει η Επιτροπή προτίμηση θεσμικά. Απλώς επιμένουμε πάντα ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζουμε τη φύση και τις εξουσίες, τη φύση του νομοθετήματος και τις εξουσίες που χρειάζονται για να θεσμοθετηθεί και βέβαια αυτό βάσει των όρων, των κριτηρίων που προβλέπει η συνθήκη. Για παραδείγματι, συμπλήρωση και τροποποίηση, δηλαδή δίνεται νέα ουσία, νέο νομοθετικό περιεχόμενο, καρονιστικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι η κατεξουδότηση πράξη και η εφαρμοτική ιστική πράξη είναι αυτή που δίνει πρακτικές ε, προδιαγραφές, πρακτικές διατυπώσεις. Αυτός ο προσδιορισμό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από αυτό θα κρυθεί και η νομιμότητα τη πράξη και η νομιμότητα του οργάνου που την υιοθετεί. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνει και να τροποποιεί ένα νομοθέτημα εάν έχει μόνο εκτελεστικές εξουσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματι, σε μία περίπτωση προσέφηκε στο δικαστήριο προκειμένου να στήσει διευκρίνηση της υπόθεσης ε, του ε, προσδιορισμού, ξέρετε, στην περίπτωση των βιοκτώνων. Επίσης, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονό ότι πολλές φορές το ζήτημα της ε, κρίσης του αν πρόκειται για κατεξοδότηση πράξη παραμένει για το τέλος των διαπραγματεύσεων εκκρεμές. Εμείς θα θέλαμε κατά τη διάρκεια των και μάλιστα και κατά την αρχή καλύτερα των διαπραγματεύσεων τουλάχιστον παράλληλα με τη συζήτηση επί της ουσίας να κρυθεί το ζήτημα αυτό γιατί στο τέλος ε, είναι στο τέλος των διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει και σε ανατροπή όλων των ισορροπιών και αναλόγως να κριθεί το αποτέλεσμα. Για το ίδιο το κείμενο τώρα θα ήθελα να πω ότι είδαμε κάποιες λεπτομέρειες την πρόταση παραδείγματι της ε, περίοδου του ενός μηνός για την επανεξέταση. Με την νέα διαδικασία της ε, επιτροπολογίας που υιοθετείται στην ε, συνήθη νομοθετική ε, διαδικασία επαναφέρουμε την επανεξέταση, δηλαδή τη δυνατότητα για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ανά πάσα στιγμή της προετοιμασίας της εφαρμοστικής εκτελεστικής πράξης να παρεμβούν Άλλωστε αυτό έκανε και το 2011 με την ευκαιρία της υιοθέτηση του Μητρώου Επιτροπολογίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν έχει τίποτα άλλο παρά να ε, επισημάνει να υποδείξει ότι προτίθεται να ασκεί στο δικαίωμα ε, εξέτασης, επίβλεψης σε ένα τέτοιο, σε μια ε, πράξη, εφαρμοστική πράξη. Άρα λοιπόν, εάν εισαγάγουμε μια διοικητική περιπλοκή, δηλαδή ένα μόνο μήνα επανεξέταση μετά τη διαδικασία της Επιτροπής, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ περιοριστικό ουσιαστικά. Περιορίζεται πολύ αυτή η δυνατότητα για επανεξέταση. Και σε όλες τι άλλες περιπτώσεις, γιατί ε, είναι λίγες περιπτώσεις που αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία, ε, πάλι η δυνατότητα είναι πολύ περιορισμένη. Και πρέπει να περιμένουμε για να υιοθετήσουμε τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και πραγματικά έχεις δίκιο ότι εκ πρώτης όψεως δεν ακούγεται τόσο συναρπαστικό αυτό. Το θέμα όμως είναι όντως σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε βασισμένοι στα προηγούμενα. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για το ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Πραγματικά πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ σωστό ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο συζητούμε αυτό το θέμα και γνωμοδοτούμε προς ε, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή, τους ε, ομιλητές, τον Chris Davis και πραγματικά ανυπομονώ να δω τις τροπολογίες σας. Προθεσμία είναι η 6η Μαΐου και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε στις 29-30 Μαΐου εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση όσοι από εσά έχετε μείνει. Σας παρακαλώ να έρθετε στην ώρα σας στις 3 το μεσημέρι για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Σας εύχομαι λοιπόν καλό μεσημέρι και καλή όρεξη.